Pronti? Prendete posto. Είστε όλοι έτοιμοι. Καθίστε παρακαλώ γιατί ξεκινάμε τις εργασίες μας. Πάμε αμέσως στο σημείο 11. Παρουσίαση ενός ενημερωτικού λεπτομερούς ε, σημειώματος για τις πιο τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το νομοσχέδιο περί Γεωργίας στις ΗΠΑ. Οπότε, συνάδελφοι, είχαμε ζητήσει μια ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία για την υιοθέτηση του νέου νομοσχεδίου περιγεωργίας στη ΣΥΠΑ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το αμερικανικό σύστημα και να το συγκρίνουμε με τη δική μας κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα αμέσως να καλωσορίσω τον Ζαν Κριστόφ Μπυρό, και να του δώσω αμέσως το λόγο. Χαιρετίζω και τους εκπροσώπους της Επιτροπής και μετά αμέσως θα γίνει η συζήτηση και ελπίζω πως οι συνάδελφοι βουλευτές θα έρθουν. Έχεις το λόγο. Ζαν Κριστόφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω τις έσχατες εξελίξεις ε, της γεωργικής νομοθεσίας των ΗΠΑ, κάνοντας ε, μια μικρή αντιπαραβολή με την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις ε, της Αμερικανικής νομοθεσίας διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις δικές μας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα εκπνεύσει σε λίγα χρόνια. Άλλα προγράμματα είναι πιο μόνιμα, αλλά πρέπει ε, το Κογκρέσο να ε, υπερψηφίσει την πρόταση χρηματοδότησης. Για να συνοψίσω, θα έλεγα ότι πολλές διατάξεις του, το, της τωρινής νομοθεσίας, σε πολλές ενισχύσεις γεωργικές συγκεκριμένα, εξέπνευσαν στις 30 Σεπτεμβρίου, ε, πρόδεκα πενθυμέρου δηλαδή, ε, και οι πληρωμές θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος του 2013 για διάφορα άλλα ε, προγράμματα, αλλά πάντως έχει εκπνεύσει το πρόγραμμα. Το επιστητιστικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο 80% μιλάμε για επιστητιστικά δελτία, τα επανομαζόμενα food stamps, ε, ανήκουν σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να επαναχρηματοδοτηθεί. Ε, εάν δεν υπερψηφιστεί η νομοθεσία για τη γεωργία, διότι το 2012 ήδη έπρεπε να έχει εγκριθεί αλλά έχει σημειωθεί καθυστέρηση και υπάρχουν πολλές παλιές ε, νομοθεσίες από το 38 και το 49 που θα εφαρμοστούν. Κάθε νομοθεσία να στέλνει την ισχύ αυτών υπό φυσιολογικές συνθήκες και φυσικά είναι παροχημένες ε, οι νομοθεσίες αυτές ε, και δεν ε, είναι λογικό να εφαρμοστούν σήμερα. Το πιο λογικό είναι παράταση κατά ένα χρόνο ενδεχομένως τη τωρινή νομοθεσία. Όμω είναι πάρα πολύ δύσκολο για δημοσιονομικού λόγου να παραταθεί το πρόγραμμα και η σχετική νομοθεσία, διότι υπάρχουν αυτόματοι σταθεροποιητικοί συντελεστέ στον προπολογισμό του που ψηφίζει το Κογκρέσο. Στο το Κογκρέσο, δηλαδή η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων, ε, νομοθετούν στον τομέα της γεωργίας ε, ε, στην ΗΠΑ. Υπάρχει πολύ μικρή επιρροή από πλευράς αμερικανικής κυβέρνησης. Τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις τους. Λοιπόν, αρχίζουμε με μια έγκριση από πλευράς του, της αντίστοιχης υπηρεσίας όπως το Κομαγκρί στη Γερουσία και στη συνέχεια περνάει από την Ολομέλεια. Η Γερουσία τον Ιούνιο ενέκρινε τη δική της ε, πρόταση για την νομοθεσία στη συνέχεια. Ε, στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει επίσης εγκριθεί η δεύτερη πρόταση, αλλά δεν έχει περάσει από την Ολομέλεια. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ε, πρέπει να εγκρίνει το νομοσχέδιο. Στη συνέχεια υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης και σύγκλησης για να φτάσει το νομοσχέδιο στον Πρόεδρο που μπορεί να προτάξει βέτο όπως έγινε το 2008 αλλά το Κογκρέσο ε, υπερπίδησε, ε, ανέρεσε αν θέλετε την αρνησικυρία του Προέδρου. Ε, ένα, μια πολύ μεγάλη τροχοπέδη στην Βουλή Αντιπροσώπων είναι ακριβώς τα δημοσιονομικά εμπόδια, συγκεκριμένα το, το μεγάλο κονδύλι για τα επισητιστικά δελτία, τα food stamps. Ε, ε, παρατηρείται συντηρητισμό σε δημοσιονομικό επίπεδο ε, και δεν είναι επιθυμητή η χρηματοδότηση, κυρίως λόγω της κρίσης. Υπάρχουν πολλά μέλη του, Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που δεν επιθυμούν περιστολή του προϋπολογισμού. Αν δούμε την πρόταση της Γερουσίας και της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Αφετέρου, διαμορφώνουμε μια σχετικά πλήρη εικόνα σε σχέση με την μελλοντική, το μελλοντικό νομοσχέδιο αν όντω εγκριθεί τους προσεχείς οι θεσμικές διαφορές ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη ακροφυγώς αναφέρθηκα σε αυτές, η εξουσία ανήκει στο Κογκρέσο, υπάρχει και ένα ε, φαινόμενο ιδιαίτερο στη ΣΥΠΑ, δηλαδή ο τρόπος εκπροσώπησης ε, στην Βουλή Αντιπροσώπων. Πρόκειται για ερετούς, για περίοδο δίαιτη, που εκλέγονται αναπεριορισμένες γεωγραφικές περιοχές και είναι σε μόνιμη προεκλογική διαδικασία ουσιαστικά. Είναι ένα άλλο μοντέλο άμεσης δημοκρατίας ε, που όμως ανοίγει το παράθυρο για ε, άσκηση ε, πίεσης από ομάδες ειδικών συμφερόντων και οδηγεί σε εξαιρετικά περίπλοκα νομοσχέδια γεωργικά διότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά συμφέροντα και πολλοί διάφοροι τους οποίους πρέπει να ικανοποιήσουν στο Κογκρέσο. Λοιπόν, 80%, 78% συγκεκριμένα του γεωργικού προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε αυτό το επιστημιστικό πρόγραμμα και με την τωρινή σημερινή κρίση σημειώνεται μεγάλη αύξηση. Δείτε το διάγραμμα, βλέπετε τις επιπτώσεις ε, της κρίσης επί του επιστημιστικού προγράμματος ε, και του προγράμματος για τα σχολεία ε, και τη διανομή τροφίμων στα σχολεία. Είναι εντάσσεται στο, πρόγραμμα, στο προνοιακό πρόγραμμα της ΕΙΠΑ, ε, αυτή η πτυχή ε, του, ε, της γεωργικής παρέμβασης, αλλά σας λέω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διοχετεύεται στο επιστημιστικό πρόγραμμα. Δεύτερο κεφάλαιο, περιβάλλον, προστασία των φυσικών πόρων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, διότι πολλά στη γεωργική νομοθεσία είναι συνάρτηση των αγοραίων τιμών, οι οποίες είναι μάλλον πλέον ε, Αυτή τη στιγμή είναι συγκυριακό το φαινόμενο κατά τη γνώμη μου. Οι πληρωμέ λοιπόν που φαίνονται εξαιρετικά σημαντικέ σε σχέση με τι άλλε ε, σχετίζονται με την προστασία του περιβαλλοντό. όμως υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, με τα κοινοτικά προγράμματα, διότι από ιστορικής πλευράς η παρέμβαση βασίζεται σε άγρανα από retirement, γιατί θεωρείται ότι ο Γιώργο έχει, ε, εμείς θεωρούμε εδώ ότι ο Γεωργός έχει έχει πολύ μεγάλη, μεγάλο ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στη ΣΥΠΑ χρησιμοποιούν τα προγράμματα αγρανάπαυσης, ούτως ώστε να διαχειρίζονται ε, τα δάνεια προς τους γεωργούς, ε, δηλαδή κάτι που προσωμιάζει με τον δεύτερο πυλώνα το δικό μας ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αν δούμε, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Τη δεκαετία του 90 ήταν πρωτοπόροι οι Αμερικανοί, πέρασαν δηλαδή στις άμεσες αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, ουδέτερες ως προς την παραγωγή, αλλά έκτοτε από το 2000 και μετά ε, ε, ε, επέστρεψαν στο παλιό σύστημα όπως στην Ευρώπη και θέσπισαν σύστημα ενισχύσεων που αποσκοπούν στην μέγιστη δυνατή προστασία των γεωργών για την μείωση του εισοδήματος, για περιπτώσεις εξηρασίας παραδείγματος χάρη ή για μη ευνοϊκές αγορές μέσα των προϊόντων Του. Είναι μάλλον περίπλοκο το σχέδιο και μάλλον αναποτελεσματικό όταν κάνουμε την ε, αντιπαραβολή με το δικό μας ε, πρόγραμμα και τις άμεσες ενισχύσεις και τους δύο πυλώνες. Εάν ε, δούμε τώρα όχι την επισητιστική πτυχή αλλά το θέμα της καθαρής στήριξης προς τους γεωργούς, ιδού ο κατάλογος των διαφόρων ενισχύσεων ε, έχουμε πάγιες αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ε, που μοιάζουν με τις δικές μας ενισχύσεις, ενιαίες τρεματικές ενισχύσεις, οι οποίες όμως βασίζονται σε ένα σύστημα πληρωμών που ξαναλέω είναι συνάρτηση των αγοραίων παγκοσμίων τιμών των προϊόντων και η κυβέρνηση καλύπτει την διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη τιμή και την αγοραία τιμή. Επίσης υπάρχουν αντικυκλικές ε, όπως λέγονται πληρωμές για να καλύψουν τη διαφορά στην τιμή λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Επίσης υπάρχει εξασφάλιση της συγκομιδής, δηλαδή οι γεωργοί δίνανται να έχουν και μια εξασφάλιση του εισοδήματος τους βάσει αυτού του συστήματος. Έχουν και συστήματα που μοιάζουν πολύ με την παλιά ε, ΚΑΠ για το γάλα και για τη ζάχαρη, η ε, δεκαετία του 80 και υπάρχουν και νέα συστήματα, δηλαδή αντισταθμητικές ε, εισοδηματικές ενισχύσεις. Άκρε, αυτό είναι το ακρονίμιο του συστήματος που που ε, αντικαθιστά τα εχέγγυα που δίνονταν, διότι το Κογκρέσο έκρινε ότι ήταν ε, υπερβολικά ε, περίπλοκο το σύστημα και το 2008 το λόμπινγκ των ασφαλιστικών εταιριών επέβαλαν ακριβώ τη διατήρηση, παράλληλη διατήρηση αυτών των δύο συστημάτων, όπερ και αναποτελεσματικότητα, ε, συγγνώμη, εξού και η αναποτελεσματικότητα του συστήματο. στη συνέχεια αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του έτου, εκτό προπολογισμού, να εκταμιευθούν ληφθούν νέα ποσά, ε, δηλαδή πιστώσεις αναλήψεις υποχρεώσεων που έγιναν από το 2000 μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο. Δηλαδή ε, προς αυξήσεις ε, στα γεωργικά κονδύλια που ψηφίστηκαν στα πλαίσια της ψηφοφορίας για τον πόλεμο στο Ιράκ παραδείγματος. Χάρη στη συνέχεια αυτά τα έκτακτα μέτρα που δεν ήταν έκτακτα γιατί επανέρχονταν συστηματικά αποφασίστηκε να γίνει ένα νομοσχέδιο, ένα σύστημα, το ΣΟΥΡ, για την κάλυψη των φυσικών φυσικών καταστροφών. Ε, είναι πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα ε, σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Αυτή τη στιγμή, εφόσον ε, το 2010 και 2011 αυξήθηκαν οι παγκόσμιε τιμέ των προϊόντων. Αυτό το πρόγραμμα των αντικυκλικών πληρωμών, τα δάνεια που δίνονται προς τους γεωργού για τη διατήρηση της παραγωγή τους σε αποθήκε συνδέονται με την ε, τωρινή κατάσταση στην αγορά και στην προσωμείωση που γίνεται για το μελλοντικό νομοσχέδιο. Το Κογκρέσο θα κάνει μια προβολή για δεκαετή περίοδο σχετικά με το κόστος ε, του προγράμματος, ε, η περίφημη baseline, δηλαδή οι τωρινέ δαπάνες του συστήματος. Και θα εξεταστεί αν θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο αυτές οι ενισχύσεις, διότι θα είναι σε καλή κατάσταση οι αγορές. Κατά τη γνώμη μου θεωρήθηκε κίνδυνο να θεωρηθεί ότι θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο οι πληρωμέ ε, και τα μέλη του Κογκρέσου, βλέποντα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, είδαν ότι στο νομοσχέδιο αυτό που κοστίζει ακριβά είναι αποσυνδεδεμένε άμεσε ενισχύσει ε, και στη συνέχεια το προπολογισμό για την ε, προστασία των φυσικών πόρων. Όμω, δημιουργούνται ψευδεστήσει. Μπορεί κάποιο να θεωρήσει ότι οι αντικυκλικέ πληρωμέ φτάνουν σε 5, 6, 7 δι αμερικανικά δολάρια ανάλογα με τις ε, συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά. Δηλαδή ε, η τεχνογνωσία τους ίσως χωλαίνει σε σχέση με αυτά που επιτυγχάνουμε εμείς εδώ με τις αξιολογήσεις αντικτύπου που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προπολογισμό τώρα για τα ε, χέγγε, για τις ασφάλειες. Τα κονδύλια αυξάνουν, καλύπτονται τα ασφάλιστρα εν μέρη από την κυβέρνηση, χρηματοδοτείται το, η λειτουργία του συστήματος με πληρωμές προς τι ασφαλιστικές εταιρείε και στη συνέχεια οι αντασφαλίσεις χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Δεν έχουμε τα στοιχεία για το 2012, αλλά έχουμε δει προσωμιώσει ε, που αναφέρουν για 16, 17 έω και 24 δι αμερικανικά δολάρια. Ε, εάν ε, δούμε πόσο κόστιζε η ασφάλεια για το 2012, 20 δις και μπορούμε Μάλλον, ε, το 2012 μπορούμε να φτάσουμε τα 20 δις, ενώ όταν θεσπίστηκε πρώτη φορά το πρόγραμμα ήταν στα 5 δις. Βλέπετε ότι είναι ισχυρότατες οι διακοιμάνσεις ε, από χρόνο σε χρόνο και ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ένα αντίστοιχο σύστημα στην Ευρώπη. Το ασφαλιστικό σύστημα έχετε ένα λεπτομερές κομμάτι της παρουσίασης που αναφέρεται σε αυτό. Εγώ είμαι ιδιαίτερα επικριτικός, διότι αν δείτε ποιο είναι το κόστος για το φορολογούμενο, και τελικά ε, ποιε είναι οι πληρωμές που λαμβάνει ο Γεωργός. Ε, βλέπουμε φοβερές απώλειες ανάμεσα στα δύο, ε, κυρίως λόγω των πληρωμών προ τι ασφαλιστικέ εταιρείε που διαχειρίζονται αυτό το σύστημα. Φαίνεται να μην είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα και προτείνονται εξοικονομήσεις και προτείνεται ένα δωρεάν για του γεωργού σύστημα που θα είχε μικρότερη κάλυψη αλλά σφαιρικά θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Πάντως, ε, το τωρινό σύστημα σίγουρα δεν είναι καλή έμπνευση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τώρα τις δύο προτάσεις ε, ε, της Γεροσίας που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια και την πρόταση της Βουλής των Αντιπροσώπων που ουσιαστικά είναι η πρόταση μόνο της Επιτροπής Γεωργίας Βουλής των Αντιπροσώπων διότι τα ποσά στα οποία καταλήγουν μέσα στην πρότασή τους, ε, δηλαδή εξοικονόμησε 10 χρόνια της τάξης των 35 δις δολαρίων ε, για την ε, γεωργική νομοθεσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση διαφέρει λίαν από την πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στα δύο. Προεδρεύει ο, ο, Πολ Ράιαν που είναι υποψήφιος και για αντιπρόεδρο αυτή την Επιτροπή επιθυμεί σοβαρή περιστολή των ε, του επιστημιστικού προγράμματο. Σε δύο περιπτώσει, είτε μιλάμε για την Επιτροπή Γεωργίας Συμβουλή Αντιπροσώπων είτε για τη Γερουσία. Ε, το δημοσιονομικό κόστο οφείλεται ακριβώ στο επιστημιστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα προστασία των φυσικών πόρων. Αυτέ οι δύο προτάσει επίση αποσκοπούν στην ε, λήξη του συστήματο αμέσων ενισχύσεων. όμω, όταν λέει στον τύπο το Κογκρέσο ότι θα καταργήσει όλε τι άμεσε ενισχύσει, δεν αληθεύει αυτό επουδενή διότι αυτό που θα ε, καταργήσουν με όλα αυτά τα προγράμματα που είδαμε είναι ε, το κομμάτι των ε, πάγιων αποσυνδεδεμένων πληρωμών, που παραδοσιακά είναι αυτό που δημιουργεί και τις λιγότερα, τα λιγότερα προβλήματα για τις τρίτες χώρες, διότι είναι το σύστημα που συνάδει σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα υπόλοιπα με τους κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπόριου. Αντίθετα, η Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων θέλουν να αναπτύξουν το ασφαλιστικό σύστημα ε, ανταυτού και το σύστημα παροχής εγγυήσεων για κάλυψη απώλειας εισοδήματος, ε, για ε, το διαφυγήν κέρδος. Δηλαδή, αν πάρουμε την πρόταση γερουσία, θέλουν να αντικαταστήσουν και τις άμεσες ενισχύσει αλλά και τις αντικυκλικές πληρώμες, καθώς και το σύστημα ΑΚΡ για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος, έχοντας ένα σύνολο που βασίζεται αφενός στις ασφάλειες και αφετέρου στη στήριξη την εισοδηματική όταν παρατηρείται μεγάλη μείωση. Η πρόταση της Δηλαδή, Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων διαφέρει ε, κατά τι. Ε, είναι μάλλον πιο περίπλοκο το σύστημα. Αλλά συνοψίζοντα, θα έλεγα ότι η γενική ιδέα είναι να καλύψουμε τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματο ε, για του γεωργού με ε, αρκετά φιλόδοξο τρόπο, διότι ενεργοποιούνται πληρωμέ ε, για απώλεια εισοδήματο μόνο του 10% ε, και σε αυτό αντιτίθεται σε μεγάλο βαθμό η πιο συντηρητική πτέρυγα των ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο να καλύψουμε τέτοιε απώλειες εισοδήματο 11% για επάγγελμα όπως αυτό του Γεωργού, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνονται τόσο έντονες συζητήσεις στην Βουλή των Αντιπροσώπων. τώρα, σε σχέση με τις ε, διεθνείς ε, πτυχές, ε, διότι με ρωτήσατε κάτι σχετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση ε, αυτή τη στιγμή οι ΙΠΑ έχουν ε, διάφορα προγράμματα, εκ των οποίων κάποια είναι ε, συμβατά με το πράσινο κουτί του ΠΟΕ, άλλα πάλι κοινοποιούνται με τρόπο ώστε να είναι συμβατά, παρότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη συμβατότητα. Αν κάνουμε προσωμιώσεις για το 2012 με την αρκετά εντυπωσιακή ομολογουμένως ξηρασία, Εάν δηλαδή βασιστούμε ε, στην υπόθεση ότι σε ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις ε, θα πληρώσει ο φορολογούμενος 17, 18 έως και 24 δις δολάρια, ο μόνος τρόπος για τις ΕΥΠΑ να συμμορφώνονται με τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις τους, δηλαδή για την αθρηστική μέτρηση ενισχύσεων, το περίφημο AMS, γιατί αυτό είναι το σύστημα του που ρυθμίζει τις άμεσες αποσυνδεδεμένες πληρωμές. Λοιπόν, είναι ένα τρόπος κοινοποίηση που όμως είναι ιδιαίτερα, που μπορεί να αμφισβητηθεί και η αυστηρή Αυστραλία, ο Καναδάς ε, ε, και όχι μόνο θεωρούν ότι αυτό το, αυτός ο τρόπος κοινοποίησης ε, αντιβαίνει στους κανόνες του ΠΟΕ. Στη συνέχεια το, η Βραζιλία συνεχίζει τις επιθέσεις της για το βαμβάκι αλλά η νομολογία του ΠΟΕ για αυτό το θέμα είναι πολύ πιο γενική από τα ειδικά προβλήματα και οι προτάσεις του Κογκρέσου σίγουρα δεν θα οδηγήσουν σε επίλυση των διαφορών, διότι ο στόχος τους είναι μάλλον να καταστήσουν τις πληρωμές ε, ακόμη περισσότερο εξαρτημένες ε, από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, παρότι αποσυνδεδεμένες ε, και άρα σε έτη χαμηλών γεωργικών εισοδημάτων και εξηρασιών ή άλλων φυσικών καταστροφών θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι με την πρόταση του Κογκρέσου το γεωργικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ θα καταστεί πιο συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ ε, ε, ε, νομίζω ότι εύκολα στο μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ενώπιον των διαιτητικών οργάνων του ΠΟΕ την συμβατότητα του γεωργικού νομοσχεδίου με τους διεθνούς κανόνες. Τώρα, σας μιλούσα για το σύστημα ασφαλίσεων και ενίσχυσης του εισοδήματος ενώ ταυτόχρονα προτείνονται περικοπές στα περιβαλλοντικά προγράμματα παρότι με τις αξιολογήσεις ε, που ε, γίνονται βλέπουμε μάλλον θετικά αποτελέσματα για τη διάβρωση εδάφους, για την ε, απώλεια της βιοπικιλότητας και συναφή ζητήματα φαίνεται ότι έχουν θετικές επιπτώσεις. Τώρα για το επιστημιστικό πρόγραμμα αληθεύει ότι είναι βελόρια τα ποσά 47 εκατομμύρια Αμερικανοί φέτος θα λάβουν τέτοια δελτία. Είναι απίστευτα υψηλός ο αριθμός. Όντω υπήρξε κατασπατάληση πόρων όπω ισχυρίζονται οι Ρεπουμπλικανοί. Όμω οι αξιολογήσει που γίνονται καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον αυτά τα προγράμματα είναι χρήσιμα ε, από κοινωνική πλευρά, ε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που χωρί αυτά τα προγράμματα θα είχαν πρόβλημα επιβίωση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης όταν ε, βλέπουμε τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του γεωργικού νομοσχεδίου ότι αν δεν, αν ε, ότι αν δεν άλλαζε τίποτα, ε, το κόστος θα ήταν 995 δις ε, και αυτό που προτείνεται τώρα από τη Γερουσία είναι μείωση 23 δισεκατομμυρίων. Η Επιτροπή Γεωργίας προτείνει μείωση 35 δισεκατομμυρίων ε, και τελικά όταν ε, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 995 δισεκατομμύρια, το επιστημιστικό πρόγραμμα καλύπτεται 772. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση στη δική μας γεωργική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατείνει ένα πρόγραμμα που εδράζεται επί των άμεσων ενισχύσεων ε, και έχω την εντύπωση ότι με τις νέες εξελίξεις ε, το αμερικανικό νομοσχέδιο θα μεταεξελιχθεί σε ένα πρόγραμμα προστασίας ε, των γεωργών το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε διεθνές επίπεδο. Από αυτή την πλευρά εμείς δείχνουμε πολύ μεγαλύτερη συνέπεια στην πολιτική που ακολουθούμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα γιατί έχουμε τον ίδιο στόχο ενώ οι ΙΠΑ καρκινοβατούν. Άλλαξαν το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων, επανήλθανε μετά ε, από πλευράς ε, διεθνούς συνεργασίας ε, και για να μην υπάρξουν επιβλαβείς επιπτώσεις για τρίτες χώρες δεν κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί. Δεν ασχολούνται από ό,τι φαίνεται στο Κογκρέσο με τον ΠΟΕΒ. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Έρευνας του Κογκρέσου που αναφέρει ότι παρά την παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του ΠΟΕ αν τελικά εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν διέπεται ε, το αμερικανικό πρόγραμμα από τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς ε, για την Ευρώπη είναι ότι ε, παρότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό το σύστημα, ε, μπορεί να προστατεύσει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς παραγωγούς και άρα θα βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση για τις εξαγωγές, διότι θα έχουν αυξημένα εισοδήματα κρατώντας χαμηλά τις τιμές τους και άρα θα είναι πιο επιθετικοί για τις εξαγωγές, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συγκριθούμε με άλλες χώρες ε, όπως η Ελβετία ε, θα λέγαμε ότι είμαστε πρωτοπόροι ως προς ε, την πειθαρχία, δηλαδή θεσπίζουμε ενισχύσεις που δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στην παγκοσμία αγορά. Χώρες όπως η Ρωσία δίνουν όλο και περισσότερο συνδεδεμένες ενισχύσεις, η Κίνα το ίδιο, η Ουκρανία το ίδιο και η Βραζιλία εξάλλου. Οι ήπα, μάλλον θα καταργήσουν ε, τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις τους και θα επαναφέρουν ε, ε, αντικυκλικά προγράμματα. Αυτό δημιουργεί ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Καλό είναι που είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε ηγετική θέση, αλλά αν δεν μας ακολουθεί κανένας, τότε ίσως να έχουμε και πρόβλημα. Ευχαριστώ. Bene, grazie. Grazie a... Ευχαριστούμε πολύ, Ζαν Κριστόφ Μπυρό. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, τα όσα μας είπες ε, έχουν προκαλέσει πολύ προβληματισμό οπότε ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση παρακαλώ τους συναδέλφους να ζητήσουν το λόγο να ε, δώσω λοιπόν το λόγο στον Άγνου και μετά στον Τόρφμαν Ευχαριστώ Πρόεδρε ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή. Νομίζω πως αναφέρατε, γιατί έχασα λίγο το μέτρημα, αναφέρατε τουλάχιστον τέσσερις τρόπους για προστασία των εισοδημάτων των γεωργών. Και αυτό καταρρύπτει το μύθο ότι οι Αμερικανοί γεωργοί δεν επιδοτούνται, που είναι κάτι το οποίο επανελειμμένως ακούω. Να σας ρωτήσω όμως ως ε, άτομο και ως άτομο που κατανοείτε αυτά τα πράγματα, εσείς προσωπικά είστε υπέρ κάποιου από αυτά τα συστήματα που περιγράψατε. Βλέπετε δηλαδή ότι κάτι από όλα αυτά ξεχωρίζει ως αποδοτικό προς τους γεωργούς, ότι είναι σχετικά εύκολο στη διαχείρισή του, ότι είναι κέριο. Μπορεί να έχετε προσωπική γνώμη γι' αυτό θα με ενδιαφέρει να την ακούσω. Αναφέρατε επίσης ένα, ένα πρόγραμμα ε, ε, Με εντυπωσίαση που άκουσα ότι συμβαίνει αυτό στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε, 200, ε, έχουμε τιμές 200 ε, δολάρια τον τόνο στο, στα σιτηρά, στο, Στάρι, με εντυπωσιάζει να ακούω κάτι τέτοιο. Στην αρχή είπατε ότι ο πρόεδρο έχει δικαίωμα αρνησικυρία, το οποίο όμω μπορεί κανεί να καταρρύψει. Εγώ νόμιζα ότι η αρνησικυρία αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανεί να το καταρρύψει. Μπορείτε να, να, να ορίσετε τι σημαίνει η λέξη βέτο στην Αμερική, στα Αμερικάνικα. Και επίση ε, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα περιγράφει τη Γεωργία ω επάγγελμα. Αν είναι κανείς όμως επαγγελματία, ε, κάνει μια υπηρεσία, προσφέρει μια υπηρεσία και τη χρεώνει. Όμως ε, οι γεωργοί στην ουσία πληρώνονται. Εμείς την γεωργία τη λέμε εμπόριο, όπου κανείς επενδύει, αναλαμβάνει κάποιο κίνδυνο. Ίσως να είναι κάπως ελαφρόμυλο αυτό, αλλά τα ακούω που και που και θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. αγνή ο Ντόρφμαν και μετά ο Μάρτιν Όσλινγκ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας για όλους. Μερικές σκέψεις, επιτρέψτε μου. Στην αξιολόγηση σας είπατε ότι ο Αμερικανικός δρόμος που είναι προσιλωμένους σε αντικυκλικές ε, πληρωμές ε, δεν είναι το σύστημα του μέλλοντος. Δεν είμαι τόσο βέβαιος γιατί βλέπω τις συζητήσεις στην Ευρώπη για το σύστημα ποτιστήρι το λέω εγώ, γιατί ανεξάρτητα από τις τιμές κάθε χρόνο ε, δίνουμε στρεματικές ενισχύσεις, έτσι μοιράζουμε σε όλους. Και υπάρχει και μεγάλη κριτική εδώ για τις εκμεταλλεύσεις που ε, φέτος θα πάνε πολύ καλά, παρόλα αυτά δίνουμε στραματική ενίσχυση. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ε, αυτές οι αντικυκλικές πληρωμές των Αμερικανών ε, δεν είναι και τόσο το θέμα του μέλλοντος. Και για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις και τις εταιρείες, τις επικρίνατε, αλλά και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρώπη και εδώ ανήκει και η Ιταλία από την οποία εγώ προέρχομαι, αλλά και η Γερμανία και η Ισπανία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν συστήματα γεωργικών ασφαλίσεων πάρα πολύ αποτελεσματικά και προσπαθούν να τα επεκτείνουν ακόμα περισσότερο. Και αυτός ο γενικός αφορισμός σας στη διαφάνεια που λέει όταν, βλάπτει όταν υπάρχει μια περιβαλλοντική καταστροφή, αυξάνουν οι τιμές. Αυτό μπορεί να ισχύσει φέτος που ήταν μεγάλη η εξηρασία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αν έχετε όμως ε, ή ε, ε, αμπέλια και τα καταστρέφει το χαλάζει, ε, δεν ε, υπάρχει στην Ευρώπη σύστημα αντιστάθμισης. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά κάτι άλλο που είπατε. Το θέμα των δελτίων σύντησης. 18 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο το υπολόγισα περίπου, που σημαίνει κατά κεφαλή 250 δολάρια ε, το χρόνο τους δίνουν δελτία για να σητίζονται οι πολίτες. Καταλαβαίνετε ε, για ποια τάξη μεγέθους μιλούμε. Είπατε ότι αυτός είναι ο Αμερικανικός δρόμος και θα οδηγήσει σε μια επιθετική παρουσία της Αμερικανικής Γεωργίας στην παγκόσμια αγορά. Δεν κατάλαβα το συλλογισμό σας πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό το σύστημα επισητιστικής βοήθειας με τα δελτία κανονικά δεν επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι εσωτερικό πρόγραμμα των ΗΠΑ. αυτό. Τι δουλειά έχουν οι, οι διεθνείς αγορές κανονικά, θα πρέπει να είναι άσχετο αυτό. Είναι μια εθνική δράση, αφορά το 20% ε, των χρημάτων που απομένουν, που είναι 20 ε, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πολύ λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε λίγο να μου το διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Χόισλινγκ. Πολύ συναρπαστικό μου φάνηκε ε, ε, αυτό. Και επίση αυτό που είπατε για την Ευρώπη, ότι όλα πάνε καλά στην Ευρώπη και οι Αμερικανοί δεν ε, εντάσσονται στον ΠΟΕ. Οι Αμερικανοί λίγο διαφορετικά τα βλέπουν. Και θα με διέφερε να μάθω και την άποψη σας, γιατί είχαμε πάει πέρυσι με την Επιτροπή Γεωργίας ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, θα, ήθελα να ακούσω την ίδια παρουσίαση από ένα Αμερικανό, <laughs> να δω πώς θα μας τα πει αυτός. Ε, δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα. Τα δύο τρίτα δίνονται για το επιστημιστικό πρόγραμμα και αυτό είναι κλασική κοινωνική πολιτική. Γιατί είναι μέσα στο γεωργικό προϋπολογισμό αυτά. Αυτό με εκπλήσει. Και ποιος έχει δικαίωμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Είναι όλοι άνεργοι, είναι στην πρόνοια. Πώ θα μοιράζουν αυτά τα δελτία σύντηση, ποιος θα δικαιούται. Και ένα άλλο που είναι πιο ενδιαφέρον για τη δική μα συζήτηση εδώ στην Ευρώπη. Το σύστημα των ασφαλίσεων οδηγεί στην αύξηση του προπολογισμού. Έχει ξεπεράσει την του πλαίσια. Ακριβώς γιατί είχαν μεγάλη ξηρασία και πρόβλημα στη συγκομιδή. Χαλάσανε οι σοδιές, καταστραφήκανε. Στη Γερμανία υπάρχει μια ασφάλιση ε, για το χαλάζι ας πούμε, αλλά αυτό το ταμείο το επομίζονται οι ίδιοι οι αγρότες, πληρώνουν, καταβάλουν εκεί κάποιες εισφορές αμοιβέ. Ε, υπάρχει ένα κρατικό πλαίσιο. Τι γίνεται όμως με τις ασφάλειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγορά τα ρυθμίζει αυτά. Και αν φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο σύστημα στο δεύτερο πυλώνα, τι θα γίνει. Τι θα γίνει αν επεκταθεί το σύστημα και οικοδομηθεί και στην Ευρώπη όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα γίνει με το δεύτερο πυλώνα αν έχουμε τέτοιου είδους γεωργικών ενισχύσεων ή προ βλημάτων θεομηνιών που καταστρέφουν τις οδιές κτλ. Ε, το σύστημα δεν είναι αρκετά υπολογίσιμο ως προς τις ε, επιπτώσεις και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ορθός δρόμος αυτός να ακολουθήσουμε και στην Ευρώπη. Το ίδιο με τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία, θα με ενδιαφέρει τι γίνεται. Τι παίρνει τελικά ο Αμερικανός αγρότης, τι φτάνει στη τσέπη του αγρότη. Ε, σε σχέση και σύγκριση με την Ευρώπη. Τελικά τις κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνει ε, ο, ο Αμερικανός αγρότης, πόσο μπορούμε να τις υπολογίσουμε σε σχέση με το συνολικό του εισόδημα, είναι αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκές. Και επειδή είναι και η προεκλογική εκστρατεία τώρα στις Ηνωμένες ε, Πολιτείες, ε, και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και κατά τη διάρκεια των εκλογών η νομοθετική εννοώ. Ε, πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις, θα μπουν περισσότερο στο δρόμο των γεωργικών ασφαλίσεων ή στην εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος. Ε, το 10% λιγότερο, ποιος θα το ε, επομιστεί οι ασφάλειες. Αυτή είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη και τα συστήματα μεταξύ τους. Jim Nicholson e Ο Jim Nicholson και μετά Schmidt. Ε, thank you very much, Chairman. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και εγώ τον κύριο Πυρό για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Κάποια από τα ζητήματα που ήθελα να ρωτήσω ε, ήδη και με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνεται τις χειρότερες ανησυχίες μας για, για υποψίες για το τι μπορεί, μπορεί να συμβαίνει. Είχα πάει και εγώ πέρυσι ε, με την Επιτροπή Γεωργίας. Κάθε φορά που ρωτά τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ασφάλειες, εκφεύγουν, δεν θέλουν να απαντήσουν. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, χρησιμοποίησατε κάποια στοιχεία, 20 δισεκατομμύρια λέτε δολάρια για το 2012. Μα είναι πολλά τα λεφτά αυτά, είναι τεράστια η στήριξη και χρησιμοποιήσατε την έκφραση, αν δεν απατώμε, παραφράζω, δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, βγάζουν λεφτά από αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι ο λόγος να επιτρέψουμε σε ασφαλιστικές εταιρείες να λειτουργούν έτσι και στην Ευρώπη, γιατί θα είναι μόνοι κερδισμένοι, όχι οι αγρότες, οι ασφάλειες. Και μήπως χρησιμοποιούν ε, τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτές ως συγκαλυμμένη επιδότηση προς τους αγρότες σε τελική ανάλυση. Ευχαριστούμε, Τζιμ, Ο κύριος Σμιτ. Και μετά ο Κύριο Σικέρσκι. Και εγώ θα είμαι σύντομο γιατί διάφορες από τι ερωτήσει που εγώ ήθελα να θέσω έχουν ήδη τεθεί και μάλιστα θα ήθελα να επενέσω τον κύριο Άγνιου μάλιστα για την ερώτησή του. Ποτέ δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά εδώ νομίζω πως στύψε διάνα. Υπάρχει κάτι από την εμπειρία των ΙΠΑ που θα θεωρούσαμε ότι είναι λογικό να κάνουμε κι εμείς. Εχθές είχαμε μια συνεδρίαση των ε, σκιωδών για τον κανονισμό περί ανάπτυξης της υπαίθρου που είπαμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημόσιο χρήμα και παρόμοια σχέδια τα οποία να είναι ανάλογα, η θέση της ομάδας μας είναι ότι πολύ γρήγορα αυτό θα μπορούσε να αποσπάσει πολλά χρήματα από την ε, γεωργική παραγωγή στην χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Και σίγουρα ούτε οι γεωργοί θα κερδίσουν ούτε οι καταναλωτές. Κάτι τέτοιο ήταν τελείως λάθος. Ίσως θα ήταν πιο καλό να είμαστε υπέρ των συνεταιρισμών, του να προωθήσουμε τους γεωργούς για να κινητοποιηθούν, ας πούμε, οι γεωργοί να φτιάξουν ε, καμιβαία κεφάλαια δικά τους, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να δαπανηθούν ε, χρήματα, ε, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει ανεύθυνες πρακτικές. Και επίσης θα ήθελα να γιατί τα νούμερα είναι τεράστια. Αλλά πάλι είναι η Στη δική μας πρόταση υπάρχει ένα περιορισμένο κονδύλι για την ανάπτυξη πέθρου. Βλέπουμε τις, ε, την πολιτική ασφάλισης να απορροφά αυτά τα χρήματα. Όμως το σύστημα το αμερικανικό, αυτά τα χρήματα διαφορετικά θα είχαν πάει στην παραγωγή, στη στήριξη μάλλον της γεωργικής παραγωγής. Είναι ένα νέο κονδύλι που δημιουργείται για να συμπληρώσει την υπάρχουσα στήριξη. Και έρχομαι έτσι στον Τζιμ Νίκολσον. Είναι αυτός μια πίσω πόρτα για να στηριχθούν οι γεωργοί ώστε να α, παρακαμφθούν οι κανόνες του ΠΟΕ. Ο κύριος Σικέρσκι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το πρόγραμμα στήριξη και το, το πρόγραμμα. Μπορείτε να μας δώσετε και, τώρα, και πάλι τα στοιχεία για το πώς κατανέμεται αυτό σε εκτάρια ή αναεκμετάλλευση ή ίσως ανακαταναλωτή, γιατί γνωρίζουμε πως είναι 320 εκατομμύρια οι πολίτες των Ε, θα θέλαμε να ξέρουμε επίσης ποιο είναι το μέσο μέγεθος μιας εκμετάλλευσης, ώστε να είναι πιο εύκολο να συγκρίνουμε το αμερικανικό με το ευρωπαϊκό σύστημα. Τώρα, δεν ξέρω αν άκουσα καλά ότι εφόσον υπάρχουν ε, απώλειες 10% τότε οι, τα προγράμματα ασφάλισης ε, πυροδοτούνται και μόνο από τη στιγμή που χαθεί το 10% της παραγωγής. Γιατί δεν είναι πολύ το 10%, είναι μια φυσιολογική διακύμαση θα έλεγα που μπορεί να οφείλεται απλά και μόνο σε κλιματικές ε, συνθήκες. Στην Ευρώπη το επιστηστικό μας πρόγραμμα είναι περίπου 500 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια κόσμος υποφελείται. Στις ΗΠΑ, αν άκουσα καλά, είναι 47 εκατομμύρια ε, ο κόσμος που υποφελείται από αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, ε, χονδρικά 50% παραπάνω. Στην Ευρώπη είναι 18%, εκεί είναι 15%. Και άλλη μια ερώτηση. Ε, ποια είναι η ανταπόκριση του ΠΟΕ, τι λέει ο ΠΟΕ αν ε, οι ΙΠΑ δεν σέβονται τους κανόνες που θεσπίζει ο ΠΟΕ οι δικοί μας ε, επίτροποι εμπορίου όταν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις πάντοτε έρχονται πίσω λέγοντας ότι ο ΠΟΕ είναι τέλειος. Διερωτώμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Οι ΙΠΑ είναι τόσο ισχυρές ε, που απλώς μπορούν να παραβαίνουν όποτε θέλουν τους κανόνες του ΠΟΕ. Και έπειτα, η στήριξη στις περιοχές της Υπέθρου προέρχεται από διαφορετικό κονδύλι, το οποίο το διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές, είναι ε, πολιτιακή αρμοδιότητα ή ομοσπονδιακή. Πώς λειτουργεί. Μάλιστα. Εγώ νομίζω πως έγιναν ήδη αρκετές παρεμβάσεις ε, και... Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει να παρέμβει. Αν όχι, θα ξαναδώσω το λόγο στον Ζαν Κριστόφ Μπυρό για να απαντήσει. Όχι, ωραία. Ζαν Κριστόφ Μπυρό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, διάφορες ερωτήσεις που αφορούν το επίπεδο στήριξης στους ε, γεωργούς ε, στις ΕΙΠΑ και περί του μύθου της χαμηλά στηριζόμενης ε, Γεωργίας. Ε, ήδη είναι πάνω από τέσσερι οι τρόποι στήριξη, ε, Είναι 7 ή 8 οι τρόποι στήριξη. Είναι ένα γεωργό ο οποίο ενισχύεται σημαντικά. Αν δούμε τη στήριξη στα εισοδήματα των μέσων γεωργών, είναι αλήθεια πω ο μέσο όρο είναι χαμηλότερο από αυτόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει περίπου το 20% τη αξία τη παραγωγή, ενώ στη ΣΥΠΑ είναι το 10%, είναι το μισό. Βέβαια, αν φτάσουμε στον Γιώργο, έχουμε ψηλότερα νούμερα από ό,τι στον, ε, στην Ευρώπη. Αν συγκρίνουμε την αξία της παραγωγής, η Ευρώπη στηρίζει περισσότερο την ευγεωργική παραγωγή. Αυτό είναι γεγονός. Όμως υπάρχουν ε, μέσα πολύ πιο ουδέτερα για τη στήριξη, με λιγότερη στρέβλωση κυρίως για τις άλλες χώρες, πιο προβλεπόμενα και διάφανα μέσα επίσης, γιατί αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές δαπάνες που είναι αρκετά χαμηλές, ε, μπορεί ξαφνικά να είναι πολύ πιο μεγάλες εάν οι τιμές πέφτουν, πέσουν χαμηλότερα, να έρθουμε ας πούμε στις τιμές του 2002-2003. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι περίπλοκο, αλλά το οποίο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο όσον αφορά την στήριξη. Με ρωτήσατε κύριε Άγνιου αν εγώ προσωπικά έχω να σας πω κάποια συμπεράσματα. Αυτό που μπορώ να σας πω για τις ασφαλίσεις και ο κύριος Ντόρφον και αυτός με ρώτησε είναι ότι σύστημα, το σύστημα το ασφαλιστικό στην Αμερική λειτουργεί πολύ άσχημα. Αν δούμε τα τελευταία χρόνια κάθε φορά που ένας γεωργός πήρε ένα δολάριο πρίμα από την ασφαλιστική του εταιρεία έχει κοστίσει αυτό για την κυβέρνηση σχεδόν δύο δολάρια. Σε ένα τέτοιο σύστημα έχουμε 50% απώλειες στο σύστημα και είναι πολύ καλύτερες οι άμεσες ενισχύσεις της Ευρώπης και έπειτα να αφήσουμε τον Γεωργό να κάνει τη δική του αυτασφάλιση ή κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά την αποτελεσματικότητα. Βέβαια, είναι δυνατόν να φανταστούμε πολύ καλύτερα συστήματα ασφάλισης στην Ευρώπη. Το καναδικό, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι καλύτερο από το αμερικανικό, γιατί είναι το προϊόν, το αμερικανικό, πολύ μεγάλης πίεσης από τις ε, ασφαλιστικές εταιρείες ε, που έχουν πολύ μεγάλα έσοδα και έχουν μεγάλη αποδοτικότητα στο σύστημα. Το κράτος στην ουσία καλύπτει ολόκληρο το κόστος αντασφάλισης και αυτό δεν είναι φυσιολογικό βεβαίως γιατί η ασφαλιστική εταιρεία δεν ρισκάρει σχεδόν τίποτα μέσα στο πλαίσιο του Αμερικανικού συστήματος. Σίγουρα λοιπόν στην Ευρώπη μπορούμε να φτιάξουμε πολύ καλύτερα συστήματα. Αυτό που έλεγα δεν ήταν επίκριση κατά των ασφαλίσεων γενικά, αλλά επίκριση κατά του συγκεκριμένου συστήματος Ε, όμως ένα σύστημα αντικυκλικών ενισχύσεων μπορεί να φέρει μεγάλη άλλες δημοσιονομικές αλλαγές και διακοιμάσεις ετησίως. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα να αυτό είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την αγρανάπαυση, το αμερικανικό πρόγραμμα Conservation Reserve Program, που είναι παλαιό και στην αρχή είχε φτιαχτεί για την καταπολέμηση της διάβρωσης και μετά έγινε περισσότερο ένα σύστημα προστασίας ε, της ε, βιοπικιλότητας, ε, βασίζεται σε μια αντίληψη ότι στην οικολογία, γιατί υπάρχουν μεγάλες συζητήσει. Ε, το ονομάζουν land sparing, εξοικονόμηση γης και όχι land sharing που είναι η μοιρασιά της γης, η κατανομή της γης ε, που είναι το δικό μας εδώ το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή αντίληψη. Land sparing σημαίνει ε, διατήρηση της γης, συντήρηση της γης. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους επιστήμονες γι' αυτό. Αν κάτι θα μπορούσε να μας εμπνεύσει είναι και αυτό το πρόγραμμα συντήρησης το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα ασφαλίσεων ε, το ανέφερα. Όσον αφορά το κόστος των επιστημιστικών προγραμμάτων, 47 εκατομμύρια Αμερικανοί ωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο είναι το πρόγραμμα των δελτίων, των επιστηστικών δελτίων. Μετά υπάρχει το πρόγραμμα στα σχολεία, η σύντηση για τις ε, ε, ανήπαντρες μητέρες. Για ιστορικούς λόγους ανήκει αυτό στο γεωργικό νομοσχέδιο ε, και για πολιτικούς λόγους, για το Κογκρέσο, το γεγονός ότι η κοινωνική ενίσχυση δίνεται μέσω του γεωργικού νομοσχεδίου επέτρεψε εδώ και 30 χρόνια να περάσουν γεωργικά και οι νόμοι με στήριξη αστικών περιοχών όπου υπήρχαν, υπάρχει μεγάλη διανομή των ε, πιστιστικών δελτίων. Η ηρωνία στην πολιτική κατάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή το ίδιο πρόγραμμα των είναι αυτό που μπλοκάρει το γεωργικό νομοσχέδιο. Έχει αντιστραφεί η κατάσταση σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή. Κατά μέσο όρο το πρόγραμμα αυτό είναι 260 με 270 δολάρια μηνιαίως που σε δελτία επισητιστικά τα οποία διανύμονται στον κόσμο. Διανέμονται στον κόσμο. Μπορούμε να αγοράσουμε μόνο λοιπόν τρόφιμα, όχι αλκοόλ, και ούτε άλλες αγορές. Είναι μια μορφή αρκετά πατερναλιστική κοινωνικής βοήθειας που όμως ε, ε, ε, γίνεται θετικά δεκτή στη ΣΥΠΑ. Δεν είμαι σίγουρος τώρα ότι δεν ξέχασα τίποτα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει νόημα στην αμερικανική εμπειρία. Τι μπορούμε να πούμε και για την αντίδραση του ΠΟΕ. Αυτές ήταν οι δυο άλλες ερωτήσεις. Το αμερικανικό πρόγραμμα έχει νόημα ως προς το ότι πραγματικά προστατεύει τον Γεωργό από τις διακοιμάνσεις. Επ' αυτού, και αυτό ήθελα να πω όταν είπα ότι καθιστά την Γεωργία τους πιο επιθετική στις εξαγωγές, δεν μιλούσα για το επιστηστικό πρόγραμμα, αλλά για αυτές τις αντικυκλικές πληρωμές, συν ασφαλίσεις, συν καταστροφές που προστατεύουν το Γεωργό, του επιτρέπουν να λάβει κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που για μια εμπορική πολιτική που είναι πολύ ευνοϊκή. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι βέβαια είναι ενισχύσει συνδεδεμένε, γιατί ευνοούν την παραγωγή, καλύπτουν ε, του κινδύνου του παραγωγού. Και κανονικά οι ΙΠΑ περιορίζονται από τον ΠΟΕ. Εσείς ρωτήσατε ποια είναι η αντίδραση του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ είναι μια γραμματεία και δεν λέει τίποτα αν κανείς δεν επιτεθεί κατά τον είπα, Μέχρι στιγμής κυρίως η Βραζιλία έχει επιτεθεί κατά των αμέσων πληρωμών, η Ένωση δεν σε έχει επιτεθεί. Αν οι προτάσεις του Κογκρέσου περάσουν, η Βραζιλία έχει ήδη πει ότι δεν θα αφήσει να γίνει αυτό χωρίς καμιά τιμωρία και η Αυστραλία εξετάζει την υπόθεση πολύ ε, προσεκτικά τώρα βέβαια οι δαπάνες του 2012 των ασφαλίσεων σίγουρα θα κοινοποιηθούν μόνο το 2015. Μέχρι να γίνει διαμαρτυρία, διαβούλευση και πάνελ θα έχουμε φτάσει γρήγορα γρήγορα στο 2018 και ίσως όλοι να το έχουν ξεχάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα της λειτουργίας του ΠΟΕ. Σας ευχαριστούμε, Ζαν Κριστόφ Μπυρό, για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση και σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προβληματισμού. Τώρα, αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις για το σημείο 11, μπορούμε να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, την ε, πρόταση τροποποίησης ε, της Επιτροπής ε, ε, ΚΟΜ 2011-625, τελικό 3 της Επιτροπής για τον κανονισμό περιθεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Παρουσίαση από πλευράς της Κομισιόν. Το Συμβούλιο θέλει να εξετάσει από κοινού αυτές τις προτάσεις, γιατί οι προτάσεις τροποποίησης της Κομισιόν για την πρόταση μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής αφορούν και οι τέσσερις την προβλεπόμενη προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από του χρόνου σε. Μόνο ένα ειδικό σημείο επιπλέον υπάρχει, το οποίο έχει εισαχθεί στην υπόθεση, στον τοσχέ για την χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση, εποπτεία της κοινή γεωργικής πολιτικής και αφορά την διαφάνεια. Η Κομισιόν προτείνει νέους κανόνες για τη δημοσίευση πληροφοριών για όλους τους δικαιούχους ε, των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Κονδυλίων, ώστε να ληφθούν υπόψη αντιρρήσεις που διατύπωσε το ΔΕΚ. Θυμίζω ότι το 10 είχε, φέρει, είχε ε, κάνει έσταση ε, όσον αφορά τη διαφάνεια περί των δικαιούχων των ενισχύσεων. Ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί στις 17 Οκτωβρίου 2012, 17 Οκτωβρίου στις 12 και είναι ανοιχτή μόνο για την τροποποίηση των διατάξεων που πρόσφατα έχουν εισαχθεί. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να ασχοληθούμε ίσως πριν από αυτή την τελευταία πτυχή διαφάνεια, με τη διαφάνεια και άρα θα δώσω αμέσως το λόγο στην Κομισιόν για μια παρουσίαση των νέων προτάσεων και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Θα έπρεπε να είναι παρόν ο Γενικός Διευθυντής Μέγκελ. Είστε παρόν, μάλιστα. Οπότε σας δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι είναι πολύ ευγνώμων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολύ γρήγορα ασχολείται με αυτή την πρόταση. 25 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα βοηθήσει σίγουρα να ενσωματωθεί με ομαλό τρόπο στη διαδικασία μεταρρύθμισης. Η πρόταση αυτή έχει και ένα ιστορικό και επιτρέψτε μου σύντομα να σας το θυμίσω. Το προηγούμενο καθεστώς ήταν στο άρθρο 44α του Δημοσιονομικού Κανονισμού για την ΚΑΠ και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διατάξεις αυτές εν μέρει ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση στοιχείων πληρωμών για φυσικά πρόσωπα διότι θεώρησε το δικαστήριο ότι οι διατάξεις αυτές δεν τηρούσαν την αρχή της αναλογικότητας. Στη συνέχεια οι αντίστοιχε πρόνοιες ε, ρυθμίστηκαν για να καλύπτουν μόνο νομικά πρόσωπα. Δηλαδή δημοσιεύονται στοιχεία πληρωμών για νομικά πρόσωπα και μόνο αυτό είναι το σημερινό καθεστώς. Μετά ε, την απόφαση του δικαστηρίου μελετήσαμε πάρα πολύ προσεκτικά ε, το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου και πάρα πολύ γρήγορα μπήκαμε σε μια διαδικασία εκπόνησης ένα νέου συστήματος με διαφάνεια για να κάνουμε διάφορα βήματα που χρειάστηκαν το χρόνο τους βέβαια. Ε, δηλαδή ένα κείμενο θέσεων με διαβούλευση για τους ενδιαφερμένους με μια σειρά ερωτήσεων. Επίσης ε, κάναμε και μια δημοσκόπηση ε, με τη μορφή του Ευρωβαρομέτρου για να δούμε τι φρονούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τη διαφάνεια. 62% λοιπόν των πολιτών ήταν υπέρ της ε, δημοσίευσης ε, στοιχείων ε, των δικαιούχων, μόνο 22% ήταν κατά λάβαμε υπόψη μας τις αποφάσεις για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου ε, το 2009 και 2010 που ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πρόταση που να επιτρέπει υψηλό βαθμό διαφάνειας και εδώ παραθέτω την ε, έκθεση και το ψήφισμά σας για την απαλλαγή το 2009 υψηλό επίπεδο διαφάνειας και επίσης λάβαμε υπόψη πάρα πολύ προσεκτικά τις διατάξεις των νέων δημοσιονομικών κανονισμού που συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο πριν το θέρος ε, στα τρία θεσμικά όργανα και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός υποθέτω ότι πολύ σύντομα θα τεθεί σε ισχύ. Τα άρθρα 56 που αφορούν τη συνδιαχείριση ζητούν μία εκ των υστέρων ε, ετήσια δημοσίευση των δικαιούχων πληρωμών από τον κοινοπολιτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 31 και το άρθρο 31 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού ε, ε, ζητεί και τη στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα με όνομα, διεύθυνση, ποσό και ε, σκοπό της πληρωμής. Έχουμε λοιπόν νέα στοιχεία από το δημοσιονομικό κανονισμό που είναι το εγκάρσιο οριζόντιο συνολικό πλαίσιο. Ε, τη βάση αυτή λοιπόν η, επί βάση αυτή η πρόταση που έχετε ενώπιον σας εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πρέπει εδώ να τονίσουμε. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν αμφισβήτησε την νομιμότητα, το γεγονό τη διαφάνεια. Απλώ ε, ζήτησε να σεβαστούμε την αρχή τη αναλογικότητα. Το είδο και ο τρόπο δηλαδή τη δημοσίευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σκοπό τον οποίο ε, εξυπηρετεί και το στόχο πολιτικά η διαφάνεια για την, Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει δημόσιος έλεγχος με την ευρύτατη έννοια των δαπανών για την κοινή γεωργική πολιτική. Άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την άποψή μας είναι και ε, το στοιχείο της απλούστευσης. Το νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε ε, επιπλέον μορφή διοικητικού και γραφειοκρατικού ε, φόρτου, ιδιαίτερα για τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών. Εδώ μιλούμε για τη δημοσίευση στοιχείων εκατομμυρίων δικαιούχων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα Άγιαξέας το 2011 αφορούσε 7,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 7,5 εκατομμύρια που θα πρέπει να δημοσιεύονται τώρα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του νέου καθεστώτος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να είναι ενιαίο, και να εφαρμόζεται ε, με τον ίδιο τρόπο για νομικά και φυσικά πρόσωπα. Μικρή εξήγηση γι' αυτό. Πολλά κράτη-μέλη μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν διάκριση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων γιατί δεν έχουν τους αυτά τα στοιχεία. Το να κάνουμε εδώ μια διαφοροποίηση θα σήμαινε επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο. Ένα δεύτερο στοιχείο. Τα, τα διάφορα στοιχεία του συστήματος είναι αντίστοιχα με το προηγούμενο με τρεις βασικές αλλαγές που έγιναν κατόπιν της αποφάσεως του δικαστηρίου για να ε, συμμορφωθούμε. Πρώτα, ε, μια αναθεωρημένη αιτιολόγηση της διαφάνειας ε, για να υπάρχει δημόσιος έλεγχος των ε, δαπανών της Ένωσης. Δεύτερον, πιο λεπτομερή ενημέρωση έχουμε αναποσό και μέσων Δηλαδή, δεν λέμε για πυλώνε πρώτο και δεύτερος πυλώνα, αλλά πόσα χρήματα πήρε ο καθένα με βάση ποιο μέτρο ε, χρηματοδότησης ποιον δικαιούχων. Και τρίτον, έχουμε βάλει ένα κατόφλι, the minimis. Κάτω από ένα ποσό δεν είναι υποχρεωτική η ε, δημοσίευση ακριβώς για να σεβόμαστε την αρχή της αναλογικότητας. Τι ορίζει λοιπόν ο κανονισμός. Ε, η δημοσίευση των δικαιούχων των κονδυλίων της ΚΑΠΗ, είναι φυσικά είτε δυναμικά πρόσωπα, θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά ε, και το status quo και να αναφέρεται και η διεύθυνσή του, ε, δηλαδή ο Δήμος και ή δυνατόν ακόμα και ο ταχυδρομικός κώδικας. Θα δημοσιεύονται τα ποσά που έχει λάβει στα διάφορα οικονομικά έτη και κατανεμημένα ε, αναμέτρο, αυτή είναι η νέα απέτηση, και στο δεύτερο πυλώνα και ε, τα εθνικά ποσά και τα κοινοτικά θα πρέπει να δημοσιεύονται για να υπάρχει συνολική εικόνα των ε, ενισχύσεων. Και τέλος θα πρέπει να, υπάρξει, να υπάρχει ενημέρωση για το είδος των μέτρων και περιγραφή των μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο αναγνώστης ε, να κατανοεί ε, περί τίνος πρόκειται και ποιο ποσό είναι και τι ε, μέτρο χρηματοδοτεί. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται σε μια μοναδική ιστοσελίδα κράτος μέλους για μια διετία. Και αυτό ισχύει, είναι κάτι που λέει ο κανονισμός τώρα. Γιατί η γιατί αυτή η πληροφορία έχει νόημα, αναγνώστης έχει κάποια ιδέα για το πώς ενισχύθηκε ένας ε, δικαιούχος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη περίοδος για να μην υπάρχει υπερβολική ε, ανάμειξη στα θεμελιώδη δικαιώματα. Βάλαμε και ένα κατόφλι λοιπόν για να σεβαστούμε την αναλογικότητα, το οποίο ε, ορίζεται ε, ανακράτος μέλος, ανάλογα με το τι θεωρεί μικρό αγρότη κάθε χώρα. Μπορεί να διαφέρει λοιπόν αυτό από χώρα σε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο που θα μπορούσαν ε, τα κράτη-μέλη να ορίσουν το 1.000 ευρώ. Δηλαδή κάτω από 1.000 ευρώ δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης. Στην περίπτωση αυτή το όνομα δεν δημοσιεύεται, αλλά δημοσιεύεται ο Δήμος ή η κοινότητα, ο τόπος διαμονής, το ποσόν το μέτρο και η ε, περιγραφή του μέτρου. Δηλαδή το μόνο που δεν δημοσιεύεται είναι το όνομα. Έτσι σεβόμαστε λοιπόν την αρχή της αναλογικότητας διατηρώντας περιορισμένο ε, τον κίνδυνο δημιουργίας υπερβολικού γραφειοκρατικού φόρτου. Ακολουθούν εφαρμοστικές ε, πράξεις ε, που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κάτι που δυστυχώς δεν μπορώ να σχολιάσω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες είναι το εξής. Ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, Προσωπικών Δεδομένων μόλις εξέδωσε μία γνωμοδότηση ε, σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Χθες έλαβα το έγγραφο αυτό, ακόμα δεν το έχω αναλύσει, αξιολογήσει, αλλά την ίδια ενημέρωση έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε λάβει και εσείς αυτό το έγγραφο και αν χρειάζεται ε, να επανέλθουμε στις συστάσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. <coughs> Τι με είστε τώρα. Ακολουθεί διαδικασία. Ε, θα πρέπει το σύστημα αυτό της διαφάνειας να συνοδεύει τη μεταρρύθμιση έτσι ώστε και τα δύο να μπορούν να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Αυτό εξασφαλίζεται από τη συμπερίληψη αυτών των κανόνων για τη διαφάνεια στο οριζόντιο πακέτο, οπότε θα τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ. Τέλος, να πω ότι οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώ επειδή είναι περίπλοκο το θέμα αυτό και με τεχνικές ψυχές, είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλε τεχνικέ ε, εξηγήσει τυχόν ε, θέλετε και η ε, Επιτροπή σα και η Γραμματεία ή οποιοδήποτε μεμονωμένο βουλευτής αν έχετε ερωτήσει, είμαστε πάντα στη διάθεσή σα για περαιτέρω διευκρινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ. Εμεί ευχαριστούμε τον ε, Διευθύντη Βέγγελ για την παρουσίαση αυτή. Επαναλαμβάνω, για όλα τα θέματα που αφορούν την ένταξη της Κροατίας δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλα ζητήματα να συζητήσουμε. Αυτό για τη διαφάνεια είναι λεπτό θέμα. Ο κύριος Τζοβάνι Λαβία δυστυχώς κολλείεται και δεν ε, μπορεί να έρθει, αλλά θα μιλήσει ο Μισελ Νταντέν αμέσω για να υπογραμμίσει αυτές τις ανησυχίες που γεννήθηκαν από το ειδικό θέμα της διαφάνειας. Ο Μισελ Νταντέν και μετά έχουμε και το Λάιον και άλλους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο Τζοβάνι Λαβία ζητάει συγγνώμη για την απουσία του και θα σας διαβιβάσω εγώ τη θέση του για τις τροπολογίες που πρόσφατα λάβατε. Ο εισηγητής διαφωνεί βαθύτατα με την πρόταση δημοσίευσης των ματεπομονίμου και της διεύθυνσης ε, των δικαιούχων στην ιστοσελίδα που θα ιδρύσουν τα κράτη-μέλη για την κοινή γεωργική πολιτική, διότι αυτό αντιβαίνει στα άρθρα 7 και 8 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφος Λαβία ε, αντιπροτείνει τη δημοσίευση των στοιχείων ε, μέσω κωδίκων ε, ad hoc. Ε, δεν χρειάζεται έτσι να τηρηθεί το κατόφλι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ και κάτω του οποίου θα πρέπει η δημοσίευση να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή θα γίνεται η ταυτοποίηση με κώδικα που δεν επιτρέπει την ανείχνευση του δικαιούχου. Έτσι διατηρεί τη διαφάνεια των ατομικών στοιχείων και προστατεύεται καλύτερα η ιδιωτική ζωή των δικαιούχων της κοινή γεωργικής πολιτικής και ε, διαφυλάσσεται η ταυτότητά τους. Ε, έτσι, ε, εφόσον ο στόχος κοινή γεωρικής πολιτικής είναι η χορήγηση των γεωρικών προϊόντων και τίποτε άλλο, θα πρέπει να προβλεφθεί αυτή η νέα διάταξη. Bene, grazie Michel, George Lyon, Martin Osling. George. Lyon. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω είναι επίμαχο το ζήτημα. Εγώ έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πώς ε, μπορούμε να δικαιολογήσουμε δύο επίπεδα διαφάνειας, ένα για τους μεγάλους ε, γεωργούς και ένα για τους μικρούς. Συγγνώμη, αν έχουμε διαφάνεια τα δημοσιεύουμε όλα. Πρέπει αυτό να είναι μια θεμελιώδης αρχή. Εγώ θα προσπαθήσω πάντως να υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Έχω μεγάλες ε, ανησυχίες για αυτή την προσπάθεια ε, κάλυψης των ε, στοιχείων μέσω ενός κώδικα. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά αυτόν τον τρόπο. Όπω ε, σωστά ε, ανέφερε ο Τζοβάνι Λαβία στο σημείο που μας διαβίβασε ο κ. Νταντά. Θέλω μία απάντηση για αυτό το θέμα. Ε, γιατί έχουμε δύο ταχύτητες, δύο διαφορετικά επίπεδα. Κάποιον τα στοιχεία θα δημοσιεύονται, κάποιον άλλον όχι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτό ακριβώ. Σα ευχαριστούμε Μάρτιν Χόισλινγκ και μετά Σμιτ. Yeah. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι και εγώ υπέρ μιας οδηγίας διαφάνειας, χωρίς εξαιρέσεις. Και χωρίς να αρχίσουμε τώρα με κώδικες να ε, κρύβουμε διάφορα πράγματα. Δεν θα ε, επιβαρύνει μόνο τα πράγματα, αλλά θα έχουμε ανθρώπους που θα προσπαθούν να σπάσουν τους κωδικούς. Μα ε, η διαφάνεια είναι δεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικέ μα συνεδριάσει είναι δημόσιε. Έχουμε πόθεν έσχε. Γιατί ο φορολογούμενο να μην ξέρει τι λεφτά δίνει στου αγρότε. Και δεν θα πρέπει να δικαιολογούμαστε ούτε να απολογούμαστε. Στη Γερμανία γίνεται πάντα συζήτηση. Και μάλιστα με μεγάλο πάθο κάθε φορά. μπορώ να εξηγήσω γιατί παίρνουν χρήματα οι αγρότε. Δεν έχω πρόβλημα. Ε, κάτι σημαντικό και αυτό είναι το αποφασιστικό στη νέα πρόταση ε, υπάρχει διαφοροποίηση στο τι ε, πληρώνεται και για ποιο λόγο. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος στην παλιά οδηγία. Η διαφοροποίηση ήταν ε, επενδυτικές ενισχύσεις, τρεματικές ενισχύσεις, περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Τώρα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και Μπορεί κανείς να πει ε, ε, με ψηλά το κεφάλι στην κοινή γνώμη, μάλιστα είμαι αγρότης, έχω κάνει τα, αυτά, για το περιβάλλον, έχω πάρει αυτή την ενίσχυση. Και ε, το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τις δαπάνες μας. Τώρα, εξαιρέσεις, ε, κρυπτογραφήσεις, όλα αυτά περιπλέκουν την κατάσταση και ε, δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι θετικός στην προσέγγιση μου. Και η ομάδα μου είναι επί της αρχής ε, και καταρχήν υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σμιθ. Μάλλον συνενετική, σε συνενετική διάθεση με Συμφωνώ με τους φιλελευθέρους τώρα. Πριν συμφωνούσαμε με τον κύριο Άγνιο. Είναι τρομακτικό αυτό. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, πραγματικά έχουμε πάρει λάθος κατεύθυνση. Είναι πρακτικά τα ζητήματα. Άκουσα τις ανησυχίες του Τζοβάνι, αλλά ε, διαφωνώ, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Καταλαβαίνω αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι προσπαθούν να βρουν ένα σύστημα ε, που να ε, λειτουργεί, αλλά μην καταλήξουμε όπως ο Κάφκα σε σύστημα που τελικά είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Όντω όλοι δικαιούνται προστασία για την ε, προσωπική του ε, ζωή. Αλλά όμω αν θέλετε να είστε δικαιούχο ε, δημοσίου χρήματο, απεκδίεστε του δικαιώματό σα. Αλλιώ πώ θα έχουμε λογοδοσία, πώ θα είναι ακέραιο το σύστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν δαπανώνται δημόσια κονδύλια πρέπει να δημοσιεύονται τα στοιχεία, πρέπει να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το κοινό. Για να βλέπουν όλοι πού πάνε τα χρήματα και τι ακριβώ έχει επιτευχθεί από για την πρακτική πλευρά του Ζητήματο, ε, ότι θέλουμε άλλο ε, σετ ε, κανόνων διαφάνεια για τα νομικά και για τα φυσικά πρόσωπα. Μα άμα δεχτούμε την ίδια την αρχή, δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε ένα ιδιαίτερα δαπανήρο και περίπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα για να έχουμε αυτό, τον, αυτή τη σαλάτα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν πρόκειται κιόλα να λειτουργήσει. Οποιοδήποτε, ξαναλέω, είναι δικαιούχο δημοσίων κονδυλίων και δαπανούνται τα χρήματα για το δημόσιο καλό, πρέπει όλα αυτά να καταγράφουν γράφονται τα στοιχεία, τελεία, τίποτα άλλο. Ο αντιπρόεδρος Σεκέρισχη και μετά ο, ο κύριος Κάπουλα Λασάντος. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι κανόνες ε, χορήγησης των ενισχύσεων είναι σαφείς για τους γεωργούς, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, ε, ενισχύσεις που δίνονται μετά από υποβολή κάποιου προγράμματος, κάποιου σχεδίου. Πριν την προσχώρηση της Πολωνίας στην Ένωση έπρεπε κανείς να υποβάλει ένα πίνακα με όλα τα στοιχεία για τα κονδύλια που λάμβανε κανείς για, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ήταν ένα πολύ καλό ε, μια πολύ καλή πρακτική. Αυτές οι ε, περιπτώσεις ε, απαιτούν τη διαφάνεια καθώς και ε, αντιστάθμιση για τις ζημιές που κανείς μπορεί να υποστεί. Είναι ενδιαφέρουσες οι προτάσεις λοιπόν και στην Πολωνία ορισμένοι γεωργοί ήταν κατά του, γεγονό, του γεγονότος ότι δεν δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Κάποιοι εδώ είχαν πει ότι όλοι τα δημόσια πρόσωπα ε, δημοσιεύουν τους μισθούς τους και τα εισοδήματά τους γιατί αυτό να μην ισχύει και για τους γεωργούς. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ο Λουίς και μετά η Μπρίτα. Πολύ σύντομα να πω, Πρόεδρε, ότι συμφωνώ με όσους υπέδειξαν την προτίμησή τους για μεγάλη διαφάνεια. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι μιλάμε για δημόσια χρήματα. Άλλο είναι να αποκαλύπτει κανείς τους ιδιωτικούς λογαριασμούς ή τη εισοδήματα ενός γεωργού ε, και άλλο είναι το να δημοσιεύει τα χρήματα που λαμβάνει από την κοινότητα. Όποιος δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, ε, θα πρέπει και να ε, μην λάβει αυτά τα, αυτά τα, αυτές τις ενισχύσεις. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Προσοχή χρειάζεται εδώ. Όπως είπε και ο κύριος Λαβία. Ε, έχουμε και το ε, θέμα των δικαιωμάτων του κάθε αγρότη προσωπικά. Καλό θα ήταν και πιο έξυπνο να κοιτάξουμε τι λέει ο επόπτης προσωπικών δεδομένων. Να το μελετήσουμε, να το διαβάσουμε. Η Κομισιόν δεν το έχει κάνει ακόμα, δηλαδή στις προτάσεις της δεν συμπεριλαμβάνεται. Είναι λογικό να ακούμε ότι όταν πληρώνουμε δημόσια κονδύλια θα πρέπει να γίνεται αυτό με διαφάνεια και να παρουσιάζεται. Αλλά όλα τα κονδύλια του προπολογισμού είναι δημόσια οικονομικά. Και τώρα αρχίζουμε από ένα μικρό τομέα από τη γεωργία σε επίπεδο προσωπικό του αγρότη για να προβοκάρω λίγο. Τι γίνεται με τους μισθούς που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφουμε τα ονόματα των υπαλλήλων της διευθύνσης τους για να πηγαίνει ε, κάθε πολίτης να ελέγχει. Και υπάρχουν και διάφορες κοινωνικές δομές σε διάφορους δήμους και κοινότητες. Στη Γερμανία το έχουμε ζήσει και έχουμε επίσης δει ότι Ε, διώκονται κιόλας, υφίστανται ηθική παρενόχληση από τον κόσμο, ε, αγρότες, τους καθίζουν στο σκαμνί για λόγους ε, κομματικούς, πολιτικούς και γίνεται πολύ μεγάλη κατάχρηση αυτής της διαφάνειας, της διάβγειας. Δηλαδή, προσοχή. Να κοιτάξουμε όλες τις πλευρές, να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και να βρούμε ένα υγιή μέσο δρόμο. Ε, να μην ε, κατονομάζουμε λέτε τους μικρούς ε, και μόνο τους μεγάλους και αυτό δεν είναι λύση. Και δεν θα αναστατώσουμε τους αγρότες, γιατί ο κόσμος δεν έχει και τη μόρφωση, ούτε τη γνώση να καταλάβει την αυτά τα στοιχεία. Και το βλέπουν ως άμεση ενίσχυση εισοδήματος που πάει στη τσέπη του αγρότη και δεν έχει καθόλου έξοδα. Αν δηλώνουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα, να καταλάβουμε και να εξηγούμε ότι δεν είναι εισόδημα, ότι δεν τσοντάρουμε ας πούμε να βγάζουν περισσότερα λεφτά οι αγρότες. Όχι, προσοχή και να σκεφτούμε. Δεν είναι τόσο μανιχαϊστικά τα πράγματα και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Μπρίτα Ραϊμέ, ε, γιατί επανέφερε μια ισορροπία σε αυτή τη συζήτηση. Εύκολα ε, αποφασίζει κάποιο να δημοσιεύσει τα στοιχεία άλλων. Εγώ θα έλεγα στο, στους βουλευτές ότι άμα υπήρχε ιστοσελίδα εδώ που να δημοσιεύει στοιχεία για τι δαπάνε και του μισθού ε, όλων των παρισταμένων, τότε θα δεχτώ και εγώ να δημοσιευτούν τα στοιχεία των γεωργών, αλλά είναι απαράδεκτο να ζητήσουμε υψηλότερο πρότυπο διαφάνεια για του Γεωργού σε σχέση με αυτό που απαιτούμε για τον τον εαυτό μας. Ε, είναι, ε, ξέρω ότι πώς δημοσιεύονται στοιχεία στι οσέλιδες, αλλά άλλο είναι να έχουμε μια ε, στοχευμένη ιστοσελίδα με συγκεκριμένες πληροφορίες για τα στοιχεία των γεωργών. Προσοχή. Δεύτερον, Χρειαζόμαστε όλο και τώρα και μια συζήτηση για το σε τι ωφελεί η διαφάνεια, για, αυτό για, ποιο, για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά. Ε, Όντω μιλάμε για δημόσια χρήματα, αλλά ε, με θεμητό τρόπο χορηγούνται αυτά τα κονδύλια στους δικαιούχου που συμμορφούνται με τις απαιτήσει. Αλλιώ πρόκειται για απάτη και για ε, εγκληματική πράξη. Δημοσιεύουμε δηλαδή τα στοιχεία αυτών που ε, σύνομα είναι δικαιούχοι. για, το κάνουμε το ίδιο για τα συστήματα πρόνοια, ε, Οπότε προτείνω να δημοσιεύουμε τα στοιχεία των πολίτων των της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας, ανεργίας, σε ξεχωριστές ιστοσελίδες, ειδικές ιστοσελίδες και να, με το ίδιο επιχείρημα ότι έτσι επικρατεί διαφάνεια. Λοιπόν, Όπω σωστά είπε η κυρία Ράιμπε και επανέφερε την ισορροπία στη συζήτηση, θα έλεγα ότι οι γεωργοί δεν πρέπει να ανησυχούν ε, γι' αυτό, διότι οι γείτονε του ε, ενδιαφέρονται περισσότερο από όλου ε, για τα στοιχεία. Δηλαδή όλοι οι περίεργοι και οι κουτσομπόλοιδε θα μπουν στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, τι κάνουμε, απομονώνουμε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα που είναι δικαιούχη. Συγγνώμη, αν ισχύει αυτό για του Γεωργού, το ίδιο ισχύει για του δικαιούχου των προνοιακών επιδομάτων στους επιτρόπους, στους βουλευτές ε, και για όλους. Και δεν ε, ισχυρίζομαι ότι πρέπει όλοι να, να μην δημοσιεύουν τα στοιχεία τους, αλλά το να έχουμε ιστοσελίδες ειδικά αφιερωμένες στη δημοσίευση στοιχείων δικαιούχων ενό συγκεκριμένου τομεί. αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Όντως το θέμα είναι πολύ λεπτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Άγνιου. Και μετά Σαρβάμα. Και εντάξει, αφού είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προέκυψε πολύ η λέξη αλληλεγγύη με δύο μορφέ. Υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στους ε, βουλευτέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν συμφωνώ τακτικά με τον Σμίθ ούτε με τον Λάιον, αλλά ήταν πολύ ευγενικοί και συμφώνησαν μαζί μου σήμερα και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπαν για τη διαφάνεια. είδαμε και ένα άλλο είδο αλληλεγγύη εδώ σήμερα οι γυναίκες έχουν ε, συγκεντρωθεί και βάλουν κατά των ανδρών. Μα τι συμβαίνει. Εγώ νομίζω πως η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική γιατί πρόκειται για σημαντικά ποσά δημόσιου χρήματος και το κοινό έχει το δικαίωμα να μαθαίνει ποιοι τα παίρνουν και αν θέλουν να μπορούν να συμβουλευτούν αυτούς τους φάκελου και να, να, να, να δουν αν τα δαπανούν σωστά. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένας λόγος, ότι δηλαδή οδηγεί στο να συζητηθεί η γεωργία. Ο, ο τύπος θέλει να ξέρει πού δίνονται αυτά τα χρήματα, οι γεωργοί μπορούν να πούνε να αυτό κάνουμε, αν εμείς δεν φυτέψουμε δεν θα έχετε να φάτε. Τώρα, μήπως όμως οι, οι, οι, οι Βρετανοί, οι φορολογούμενοι πληρώνουν πολλά λεφτά για γεωργούς σε άλλες χώρες που έχουν το δικαίωμα να το ξέρουν. Να πω και κάτι σαν Βρετανός, έτσι. Ναι, Σαρβάμα και μετά και ο Σμιτ και πάλι. Ο Σμιθ. Κυρίες και κύριοι, εγώ θέλω να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα για το τι συζητάμε αυτή τη στιγμή εδώ. Προσπαθώ να μείνω ήρεμος και cool και να δείξω κατανόηση. Καταλαβαίνω τα όσα λένε οι συνάδελφοι. Όμως στη Φιλανδία οι άντρες, ο άντρας, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες ε, της Ευρώπης και ίσως και ο πλουσιότερος άνθρωπος ε, στη Σκανδιναβία τουλάχιστον στην Φιλανδία, ε, είναι στους ε, τίτλους των εφημερίδων, κυρίως των σκανδαλοθυρικών, κάθε χρόνο λέγοντας ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, παραλήπτες γεωργικής ενίσχυσης στη Φιλανδία. Και δεν έχω δει να πάει κανείς ε, να μαζευτεί εκεί λαός και να του κάψουν τη φάρμα του. Αυτό που λέω είναι ότι δεν θα πρέπει να εντοπίζουμε την ίδια τη διαφάνεια για όλα και να την έχουμε σε καραμέλα. Η διαφάνεια είναι σαν τον αέρα που αναπνέουμε ή έτσι θα έπρεπε να είναι. Και ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Άγνιου, μακροπρόθεσμα πιστεύω, ότι θα, θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αλλά σίγουρα αυτό θα δώσει λαβή για συζήτηση και μετά εξαρτάται από εμά. Να υπερασπιστούν τι κάνουν. Όσο και αν σέβομαι τον Τζοβάνι και φυσικά αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα ούτως ή άλλως, θα πρέπει να πω ότι ναι, εγώ συμφωνώ με τους άντρες σήμερα. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιθ ζήτησε και πάλι το λόγο και μετά η αντιπρόεδρος Πόλσεν. Πρόεδρε, εγώ θα μείνω έξω από την πολιτική περιφύλων του κυρίου Άγνιου, ε, αλλά θέλω να επανέλθω γιατί αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αφήνουμε ένα, μια πολύ ξεκάθαρη συζήτηση να μπει σε χωράφια άλλα. Δεν μιλάμε για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, δεν μιλάμε για τη ζωή των γεωργών, δεν μιλάμε για κοινωνικά επιδόματα. Μιλάμε για την ακαιρεότητα ε, στα μάτια του κοινού, για το τι θέλουν να πετύχουν οι γεωργικές ενισχύσεις και τι τελικά αποδίδουν και είμαστε διστακτικοί για το πώς καλά δίνει η γεωρική πολιτική και είναι η γεωρική πολιτική και αυτό γιατί υπάρχει ένας βαθμός μια κρυψίνια. Δηλαδή, ναι, είναι η γεωργική πολιτική, τα καταφέρνει καλά, δεν σας πούμε ποιος το κάνει και με πόσα. Ε, εφόσον θέλουμε να πούμε ότι είναι αποτελεσματική, μπορούμε να πούμε και ποιο την κάνει και γιατί. Ε, να πούμε αυτά συμβαίνουν στι φάρμε, αυτά συμβαίνουν για τη βιοπικιλία, αυτά συμβαίνουν που παράγουμε. Και ε, Είμαστε επιθετικοί γιατί επικρατεί μια μυστικότητα σε λάθος επίπεδο. Η Αντιπρόεδρος Πόλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω στον κύριο Άγνιου ότι ε, εγώ είμαι γυναίκα. Ε, ίσως δεν φαίνομαι γιατί είμαι ηλικιωμένη, αλλά ξέρετε έχω δέκα παιδιά, εγγόνια, δισέγγωνα, έχω και ένα τρισέγγωνο. Τέλος πάντων. Ε, εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της Ευρώπης όπου σχεδόν όλα, όλα είναι διαφανή. Ε, και μας ικανοποιεί αυτό το σύστημα. Οι γείτονε μπορούν να μπουν μέσα στον υπολογιστή και να μάθουν όχι μόνο πόσα βγάζω, πόσα έχω στην τράπεζα, πόσους φόρους πληρώνω, με ποιον είμαι παντρεμένη, πόσα παιδιά έχω, όλα τα πάντα, όλα είναι ε, δημοσιευμένα βάσει του σουηδικού συστήματος. Όταν λοιπόν ε, μιλούμε για εξέβρεση συμβαστική λύση ε, και από όσα άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική ε, δημοσίευση ε, που εξηγεί όμως για ποιο λόγο έχει λάβει ο δικαιούχος την ε, πληρωμή. Εάν είναι άμεση η στήριξη του εισοδήματος αντί να πληρώνουμε τους γεωργούς για αυτά που έχουν κάνει. Δηλαδή πρόκειται για πληρωμή υπηρεσιών και όχι για επιδόματα. Ε, δεν πρέπει να μιλάμε για επιδόματα, διότι πρόκειται για καταβολή πληρωμής για προσφορά υπηρεσιών που είναι ζωτική σημασία για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για τη δημοσίευση των στοιχείων, πρόκειται για τον τρόπο της δημοσίευσης. Ε, και νομίζω ότι είναι δυνατό να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση, δηλαδή τι ακριβώς θα δημοσιεύσουμε και με ποιο τρόπο θα το δημοσιεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Πόλσον. Ο Μισελ Νταντά τώρα. Ε, ε, τώρα μιλάω εξ ονόματός μου και όχι του Τζοβάνι Λαβία ε, σε σχέση με τις ανταλλαγές που έγιναν σήμερα. Κοιτάξτε, πρέπει να επανέλθουμε στο σημείο εκκίνησης πριν από 50 χρόνια, όταν φτιάξαμε την κοινή γεωργική πολιτική, συλλογικά κάναμε την επιλογή να μην αφήσουμε ο καταναλωτής να πληρώνει ε, τα προϊόντα στην πραγματική του ε, τιμή. Και η ενίσχυση προς τους γεωργούς είναι πρωτίστως ε, η αντιστάθμιση της υποπληρωμής του καταναλωτή. Αυτό που δεν πληρώνει ο καταναλωτής το πληρώνουν οι φόροι και πληρώνεται μέσω των άμεσων ενισχύσεων. Τα κατάλαβα όλα αυτά που είπατε για διαφάνεια και σίγουρα δεν είμαι ενάντιο. Όμω το πρόβλημα είναι υπό ποιου όρου ε, ε, επιδιώκουμε τη διαφάνεια. Αν ανεπεξέργαστα δημοσιεύσουμε αυτά τα στοιχεία, τι θα γίνει. Αν συγκρίνουμε την πραγματικότητα που επικρατεί στην εκμετάλλευση με ένα μη επεξεργασμένο στατιστικό στοιχείο, θα δείτε ότι αν κοιτάξετε αναδρομικά, ε, φτάνουν το 110-120% του πραγματικού γεωργικού εισοδήματο αυτέ οι ενισχύσει. Αν τα δημοσιεύσουμε έτσι τα στοιχεία, χωρί όμω να δώσουμε στοιχεία για το την άλλη πτυχή, δηλαδή το πραγματικό εισόδημα, ε, δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρω ότι ο, ο τύπος ε, θέλει να ασχολείται με αυτό το ζήτημα, από ποια ποσά πήρε ποιο και για ποιο λόγο. Αλλά αν ε, γίνει έτσι η δημοσίευση, θα ε, δυσχεράνουμε ε, έτσι περαιτέρω τη ζωή των Γιώργων. Εγώ ήμουν εισηγητή στο προηγούμενο εξάμεινο για την ΚΑΠΕ και πήγα σε διάφορα κράτη-μέλη και παντού οι Γεωργοί το ίδιο έλεγαν. Δεν θέλουμε επιδοτήσει, τι τιμέ θέλουμε, εγγυημένε τιμέ. Το να δημοσιεύουμε τώρα τα ποσά των ενισχύσεων, ανεπεξέργαστα, ξαναλέω, αυτό θα ενισχύσει ενισχύσει το ε, αίσθημα ενοχή ε, των ε, γεωργών. Αν θέλουμε τώρα να παρακινήσουμε τους νέους να εισέλθουν στο επάγγελμα, γιατί είναι ένας από τους δεδηλωμένους στόχους της νέας εκάπε, θα πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, ε, συνοψίζοντας, δεν είμαι κατά της διαφάνειας, αλλά πρέπει να ε, μην είναι ε, ο, ο μη και ανεπεξέργαστη αυτή η διαφάνεια. Ευχαριστούμε, Μισελ. Σερβάμα πάλι. Σύντομα, εγώ νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα του Μισελ Νταντέν και της Μαρή Πόλσον και να ε, προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το είδος στη συμβιβαστική, όπου να υπάρχουν, ε, ώστε να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να ε, δημοσιευμένες για να μπορούμε να αναλύσουμε περί τίνος πράγματος μιλάμε ευχαριστώ και εγώ θέλω να πω δύο λόγια για αυτό το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τη διαφάνεια, όπως πιστεύω όλοι μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θέλουμε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και το ίδιο νομίζω θέλει και ο Τζοβάνι Λαβία. Το θέμα είναι να μην μετατραπεί αυτή η δίκαιη επιθυμία και το βήμα μπροστά προς την αδιαφάνεια σε ένα κίνδυνο καταγραφή σε όλους τους τοπικούς, στις τοπικές εφημερίδες με το όνομα, επίθετο και διεύθυνση των δικαιούχων της ε, ενίσχυσης. Μπορεί σε ορισμένες περιοχές να δημιουργήσει δυσκολίες. Το θέμα είναι να βρούμε σωστή ισορροπία, να αποφευχθούν οι καταχρήσεις αυτή τη διαφάνεια που για σκοπούς δηλαδή όχι γνώσης των νούμερων αλλά για άλλους σκοπούς. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε και με τη βοήθεια της Επιτροπής θα δούμε ποια ισορροπημένη λύση θα μπορέσουμε να βρούμε. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και ο, κύριο, ο Διευθυντής θέλει να επανέλθει. Ναι, μισό λεπτό, George Λάιον ένα λεπτό και μετά εσείς. Μια σύντομη ερώτηση, δεν είναι γνώμη κάτι, αλλά αφού διάβασα την απόφαση του ΔΕΚ, διερωτώ με αν η Κομισιόν μπορεί να μας εξηγήσει αν πιστεύει πως αυτό θα μπορούσε να σταθεί στο ΔΕΚ και να σταθεί απέναντι σε αυτή την απόφαση. Γιατί διαβάζοντα αυτή την απόφαση δεν είμαι πεπισμένο ότι, ότι όντω ανταποκρίνεται στα θέματα που έχει θίξει το ΔΕΚ. Θέλω να ακούσω λοιπόν την άποψη τη Κομισιόν για το κατά πόσο πιστεύει ότι ανταποκρίνεται στην τελευταία απόφαση του ΔΕΚ με αυτή την πρόταση. Ναι, είναι σημαντική η ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέγελ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε μια σειρά από ερωτήσεις που έγινα. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν ξεκινούμε από μηδενική βάση. Η δημοσίευση των στοιχείων πληρωμών άρχισε το 2009 και το 2010 και το έχουν ήδη κάνει τα κράτη-μέλη δύο φορές. Ε, έχουμε εμπειρία, έχουμε ενημέρωση για τις συνέπειες αυτής της διαφάνειας. Την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα μετά τη δημοψήφιση γίνεται φασαρία στον τύπο για τις πιο ε, υψηλέ πληρωμές, για τους μικρούς αγρότες ούτε λόγος και μετά ηρεμεί και πάλι η συζήτηση και σταματά εκεί. Ε, διαβουλευθήκαμε με τους ενδιαφερομένους, μας είπαν ποιες είναι οι μεγάλες δυσκολίες και ε, τα προβλήματα που τους δημιούργησαν, ας πούμε, ο φθόνος και μόνο που δημιουργεί αυτό το καθεστώς δημιούργησε προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν εμπειρία πρώτερη και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το γεγονός ότι κάνουμε αυτή την πρόταση είναι απλό από που απορρέει. Μια απόφαση του ΔΕΚ που ε, κήρυξε άκυρη εν μέρη την προηγούμενη ρύθμιση διότι παραβίαζε το δικαίωμα προστασίας των, δεδομένων, ε, των προσωπικών δεδομένων με βάση το, της χάρτας. Ο νομοθέτης δηλαδή δεν είχε δείξει ρητά ότι είχε εξετάσει επαρκώς ε, τα διάφορα ενδεχόμενα που ε, παραβίαζαν την προσωπική ζωή με λιγότερο έντονο τρόπο. Δηλαδή αυτό που μας είπε είναι να το μελετήσουμε περισσότερο το θέμα, να μελετήσουμε διάφορες ε, επιλογές και επίσης να δούμε και ποια είναι τα ζητήματα που ε, αναφέρονται ρητά στην απόφαση. Δηλαδή ε, τι διαφοροποίηση μπορεί να γίνεται αναλογό με τα ποσά, σας ανέφερα ένα κατόφλι. Αυτό είναι ο λόγος. Και άλλη διαφοροποίηση θα μπορούσε να αφορά ειδικά συγκεκριμένους τρόπους που συνδέονται με τη συχνότητα των πληρωμών, ε, με την ε, φύση των πληρωμών, με την ουσία των πληρωμών κτλ. Αν κοιτάξετε την πρόταση θα τα ξαναβρείτε όλα αυτά. Υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό όπου εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικροί αγρότες. Εμείς επιλέξαμε ένα κατόφλι ως αντικειμενικό και ε, αν εγκριθεί μπορεί να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία για τις άμεσες ενισχύσεις για το καθεστώς για τους μικρούς αγρότες. Αυτή λοιπόν η απόφαση ε, που προτείνουμε είναι άμεση ε, απόρρια και ανταπόκριση στην απόφαση του δικαστηρίου. Γνωρίζουμε ότι το νέο καθεστώς ευσταθεί σε δικαστήριο ακριβώς γιατί έρχεται να απαντήσει στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου. Θα ήθελα να διευκρινίσω ένα σημείο Ίσως να μην το είπα με μεγάλη σαφήνεια. Εμείς δεν κάνουμε διάκριση στα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων. Καλύπτει η πρότασή μας και τα δύο, γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει από χρόν λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων. Και επιπλέον θα ήταν και πάρα πολύ ε, περίπλοκο ε, για τα κράτη-μέλη να έχουν άλλα νομικά κριτήρια για τα νομικά και άλλα για τα φυσικά πρόσωπα. Κάτι άλλο, νομίζω η κυρία Ράιμες το είπε, ε, ήταν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση ε, το σκοπό των πληρωμών ε, και των ενισχύσεων. Το είπαν και άλλα μέλη της Επιτροπής. Μα αυτό ορίζεται σαφέστατα στην πρόταση. Η πρόταση λέγει ότι τα ποσά δημοσιεύονται και συνοδεύονται ε, από εξηγήσει και για το είδος και για το, την ουσία των μέτρων που στο μέλλον θα επιτρέπουν στο φορολογούμενο να κοιτάζει τον κατάλογο, να βλέπει ποια μέτρα ε, δικαιολογούν ποιες πληρωμές σε ποιους αγρότες και όλα αυτά θα μπορεί να τα διαπιστώνει και να κατανοεί περί τίνος πρόκειται σε αυτή την πληρωμή. Ο κύριος Νταντένα, αν δεν με πρότεινε να μην δημοσιεύονται έτσι χωρίς επεξεργασία τα στοιχεία, αλλά να υπάρχει και η επιμέρους κατανομή τους. Αυτό θα μπορούσαμε θεωρητικά να το κοιτάξουμε, αλλά θα απαντήσω ότι σημαίνει ε, γραφειοκρατικό άχθος για τα κράτη-μέλη που θα το επομιστούν, οπότε θα είναι αδύνατο να δημοσιεύονται. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε και τα έχουμε με ε, σαφήνεια ε, είναι οι ενισχύσει πληρωμές. Η επεξεργασία χρειάζεται οικονομικούς υπολογισμούς, ε, μπορεί να προσβληθεί. Ε, σας είπα πόσα εκατομμύρια αγροτών. Μόνο για το σύστημα ΑΕΑΣ ήταν 7,5 εκατομμύρια αγρότες αυτοί που έλαβαν την ενίσχυση, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφεκτα αυτά τα πράγματα. Το θέμα του συστήματος ποιο είναι. Να μαθαίνει ο φορολογούμενος το ποσό που έχει καταβληθεί, ε, αυτά γνωρίζουμε και αυτά μπορούν να δημοσιεύουν τα κράτη-μέλη χωρίς να χρειαστεί να μπλέκουν τώρα με την ε, ουσία και να επεξεργάζονται τα στοιχεία. Ένα τελευταίο για να κλείσω που δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Πριν από λίγους μήνες, στα πλαίσια της συζήτησης για το δημοσιονομικό κανονισμό, το κοινοβούλιο σας ενέκρινε ένα κείμενο που περιλαμβάνει πολύ σαφή δέσμευση και προσήλωση στην αρχή της διαφάνειας και ε, τη δημοσίευση των στοιχείων ενισχύσεων, όχι μόνο της γεωργίας. Μην νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για το γεωργικό τομέα. Ε, ε, υπάρχουν και άλλες ενισχύσεις, πληρωμές ε, στην άμεση διαχείριση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έμεση διαχείριση ή ακόμα και ε, διαρθωτικά ταμεία, μια σειρά θεμάτων που έχουν όλα τις ιδιαιτερότητές τους. Δεν είναι κάτι λοιπόν που εξαιρεί τους αγρότες από τους υπόλοιπους δικαιούχους ε, κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό που προσπαθούμε είναι να βρούμε ένα ε, πρόσφορο σύστημα, ένα κατάλληλο σύστημα. Αυτό προσπαθούμε να προτείνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό περίπτωση. Για να καταλάβει ο φορολογούμενος περί τίνος πρόκειται. Με δύο λόγια. Νομίζω συμμορφούμαστε. Με το χάρη θεμελιωδών δικαιωμάτων Κατά τα άλλα το ίδιο λέει και ο επόπτης, έτσι, προστασίας πολιτικών, ε, προσωπικών δεδομένων, συγγνώμη. Ε, και θα το συμπεριλάβουμε αυτό στην πρότασή μας. Είμαστε λοιπόν προσιλωμένοι στην αρχή της διαφάνειας και ταυτόχρονα σεβόμαστε τα ε, μεμονωμένα δικαιώματα των δικαιούχων που μπορούν και να τα επικαλεστούν. Ευχαριστώ πολύ. Va ευχαριστούμε. Θα έλεγα ότι Έχουμε εξαντλήσει το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ο, ο κύριος Διευθυντής θέλει γρήγορα να πάρει το λόγο για να προσθέσει κάποιε πληροφορίε όσον αφορά την Κροατία. Γιατί εκεί θα γίνει συζήτηση. Αλλά αν θέλετε σύντομα να μας ενημερώσετε. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σημεία 10, 11, 12 αφορούν αυτή την πτυχή. Τη διεύρυνση της Ένωσης στην Κροατία και βέβαια την προσαρμογή των νομοθετικών προτάσεων της, ε, της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, το δεύτερο σημείο, το οποίο καλύπτεται από τον οριζόντιο κανονισμό που μόλις συζητούσαμε υπό την πτυχή της διαφάνειας, αλλά και σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν κάνει οι Επίτροποι για την στις άμεσες πληρωμές και για την ενιαία ε, ενίσχυση. Όπως ξέρετε όλα αυτά, ε, μάλλον το πρόγραμμα που ισχύει ε, λίγη εκπνέει το 2013 και γι' αυτό τον Ιούλιο υιοθετήσαμε μια πρόταση για τροποποίηση των δημοσιονομικών κονδυλίων μόλις θα μπει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε πω έπρεπε να μετατροποποιηθούν οι προτάσει για την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική, γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνο να αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση αυτή, ενώ οι απαραίτητε τροποποίησει για την ε, ένταξη τη Κροατία που ξεκινά 1η Ιουλίου 2013 δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτούς τους κανονισμούς περί μεταρρύθμισης. Αυτό είναι το ιστορικό της πρότασης. Η προσαρμογή που αυτή είναι βασικά τεχνική. Δεν χρειάζονται πολιτικές αλλαγές. Ε, απλώς μεταφράζεται το αποτέλεσμα των δεξιακών διαπραγματεύσεων στις προτάσεις και προσαρμόζονται κάποιες πτυχές της ε, πρότασης της μεταρρύθμισης γιατί, ε, που οφείλονται μόνο στο ότι η Κροατία θα γίνει μέλος της Ένωσης. Όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγορά, και εκεί δεν νομίζω ότι χρειάζονται εξηγήσει. Θα προχωρήσω κατευθείαν στην ε, ανάπτυξη συμπέθρου. Ε, εδώ μιλάμε για τα CNDP ή top-ups, όπως τα λέμε. Η Κροατία θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει χρήματα της ανάπτυξης πέθρου για την ε, ε, χρηματοδότηση των CNDPs, που είναι οι συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις που πρέπει να καλύψουν το κενό ανάμεσα στο φάση phasing in, ε, μέχρι ότου δηλαδή να φτάσει στο επίπεδο των 27. Η δεύτερη τιτηρότητα όσον αφορά την ανάπτυξη πέθρου σχετίζεται με την ε, θελοντική διακύμαση και τη μεταφορά μη δαπανημένων κονδυλίων που είναι και πάλι τεχνικό ζήτημα που καλύπτεται. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, ε, η κρατία ήδη έχει δεχτεί να συμμετέχει κατευθείαν στο σύστημα SPS των ενίων ε, πληρωμών, δεν θα πάει στο SAPS και ε, σχετίζεται η πρόταση αυτή με τον ε, μηχανισμό phasing in. θα ξεκινήσει το επίπεδο 25, σε επίπεδο 25% και σταδιακά θα αυξηθεί μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της Ένωσης. Υπάρχουν επίσης κάποιες προσαρμογές που χρειάζονται για τις ε, συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις. Η Κροατία θα το κάνει αυτό. Εμείς επιτρέπουμε να χρηματοδοτηθούν αυτά ε, κάποια κομμάτια αυτού από την, ε, τα χρήματα για την ανάπτυξη πέθρου. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν ε, την ε, εξουδετερώση ναρκών, γιατί η Κροατία, όπως ξέρετε, δεκαετία του 90 συμμετείχε στις μάχες των Βαλκανίων και υπάρχουν ε, γεωργικές περιοχές που είναι ναρκοθετημένες και διαρκώς γίνεται εξουδετερώση ναρκών. Ε, αυτό σημαίνει ότι καθώς περνά ο καιρός, ε, οι περιοχές αυτές θα μπορούν να μπουν και πάλι σε γεωργική χρήση και γι' αυτό χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των εκταρίων και των δικαιωμάτων που μπορεί να ε, έχουν αυτές οι περιοχές, οι γεωργικές περιοχές. 9,6 εκατομμύρια ευρώ έχουν μπει στην άκρη για να χρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες ανάγκες ως αποτέλεσμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τέλος, να πω δύο λόγια για την ε, οικονομική δήλωση για τις ενημερωμένες ε, προτάσεις για την κοινή γεωργική πολιτική ε, Φυσικά χρειάζεται ενημέρωση των δημοσιονομικών δηλώσεων. Απλώς αντικατοπτρίζονται εδώ οι προτάσεις του νέου ΜΕΦΕΦ PDP ε, που συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη για την Κροατία το 2013. Η Κομισιόν θα πω ότι φυσικά είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω τεχνικές επεξηγήσεις για την πρόταση αυτή Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν υπάρχουν αλλαγές ουσίας στις προτάσεις της μεταρρύθμισης της Κομισιόν, ούτε όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό η προσαρμογή, γιατί η Κροατία είναι τεχνικής φύσης, όπου οι αντίστοιχες απαιτήσει υπό τις πράξεις ένταξης έχουν απλώς μεταγραφεί μέσα στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ ε, Διευθυντά Μάγκελ, δεν νομίζω πως υπάρχουν παρεμβάσεις εδώ όσον αφορά την Κροατία. Οπότε ολοκληρώνεται έτσι και το σημείο της σημερινής διάταξης αυτό που ήταν το τελευταίο για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρία τη επιτροπή μας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 και 6 Νοεμβρίου για την επόμενη μας συνεδρίαση. Θα ζητήσω ωστόσο και πάλι στους συντονιστέ να μείνουν 10 λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε τα όσα δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε σήμερα το πρωί. Τέλος τη συνεδρίασης. Ευχαριστώ.